So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir sollten dennoch anfangen, auch wenn die Reihen noch Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να ξεκινήσουμε παρότι δεν είναι γεμάτα τα έδρανα. Noch ändern. Ελπίζω θα αλλάξει αυτό. Θα ήθελα να σας ε, καλωσορίσω στην ε, απογευματινή μας συνεδρίαση, η οποία ε, Στα μεγαλύτερο μέρος της είναι, αφορά μια, την ακρόαση για την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, νεολαία. Ε, υπάρχει και μια έκθεση για την ε, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την νεότητα. πελαμβάνει συστάσεις ε, την περίοδο μέχρι το 2020 και συστάσεις για μετά το 2020. Ε, η έκθεση θα παρουσιαστεί το Φεβρουάριο και αφορά τις ε, βελτιώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα ενδιαφέροντα και στόχοι των νέων, δηλαδή πώς μπορεί να υπάρξει ένα καλύτερο benchmarking ούτως σε ευρωπαϊκό αλλά και περιφερειακό επίπεδο να υπάρξει μια στοχευμένη πολιτική για την νεολαία που να είναι επιστημονικά, που να είναι τεκμηριωμένη και να διατυπωθεί συμπεριλαμβάνοντας τους νέους, τους ίδιους νέους και τις δικές τους απόψεις. Σήμερα έχουμε προσκαλέσει κάποιους ε, ομιλητές που θέλω να σας παρουσιάσω. Η κυρία Μαργκερίτ Πρωτά, ε, διευθύντρια για στρατηγική εταιρική σχέση και χρηματοδότηση α, της Παγκόσμιας Οργάνωσης της, ε, του Κινήματος των Προσκόπων, η κυρία Βίλ Μαϊαμά από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Νεολαία. Ε, συχνά εκπροσωπείται στις ακροάσεις μας το φόρουμ αυτό. Μετά ο Ντένις Ιτάσο, ο οποίος είναι βολευτής στο Συμβούλιο της, ε, του Σαν Σεμπαστιάν στην Ισπανία για πολιτισμό, τουρισμό, νεότητα, αθλητισμό και συνεργασία. Και επίσης η κυρία Τσάμπα Μπορμπόλη ε, που είναι υπεύθυνη για τον ε, διαρθωμένο διάλογο Ε, συγγνώμη, ήταν η, Λίλια, κυρία Λίλια Ελέγκοβα, η οποία ήταν στο φόρουμ των νέων στη Βουλγαρία και ο κύριος ε, Τσάμπα Μπορμπόλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών και θα ήθελα να σας αναφέρω, να σας προτείνω μάλλον μια ε, αλλαγή στη διαδικασία για να είναι πιο ζωντανή η ανταλλαγή απόψεων. Ο κάθε ένας από τους προσκεκλημένους μας θα λάβει για 10 λεπτά το λόγο για μια ομιλία και στη συνέχεια θα κάνουμε ένα ping pong, Δηλαδή θα παρεμβάλλουμε κάθε φορά ένα γύρο ερωτήσεων. Ένα λεπτό θα είναι κάθε ερώτηση, χωρίς statements, για να δίδεται άμεσα η απάντηση και να υπάρχει η δυνατότητα για μια δεύτερη ερώτηση εφόσον υπάρχει ανάγκη, δηλαδή να υπάρχει πιο διαλογική μορφή στην ανταλλαγή αυτή των απόψεων, να είναι πιο ζωντανός ο διάλογος από ό,τι μέχρι τώρα. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Ποτά για την παρουσίασή της Παρακαλώ να τηρήσετε το χρόνο των 10 λεπτών. Έχετε το λόγο, κυρία Ποτά. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Εκπροσωπώ την παγκόσμια οργάνωση του προσκοπικού κινήματος. Μιλάμε για 15 εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο, πάνω από 160 χώρες και στην Ευρώπη είμαστε κοντά στα 2 εκατομμύρια νέους ανθρώπους που είναι μέλη Είμαστε μια οργάνωση νέων, ανοιχτή προς όλους, ε, από όπου και αν προέρχονται, όποιο και αν είναι το θρησκευτικό τους, ε, ε, το θρησκευμά τους. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα εργαλείο εδώ, το οποίο να δίνει δύναμη στους νέους. Θέλουμε να δεσμεύονται, ή να συμμετέχουν ε, στις διαδικασίες, στη λήψη αποφάσεων και θα αναφερθώ επίσης τον ρόλο των οργανώσεων νεολαία στη στρατηγική αυτή. Πρώτα απ' όλα, η Ευρωπαϊκή Στρατηγική είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για τη δημιουργία μιας συμμετοχής των νέων. Μια μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων. Αυτό είναι βασικό στόχο τη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω ξέρετε, ο θελοντισμό είναι ένας πολύ καλός τρόπος της ενίσχυσης της συμμετοχής των νέων και της ενεργής συμμετοχής τους ως πολίτες. Είναι πολύ σημαντικό να νιώθουν ότι είναι μέλη μιας κοινότητας και ότι συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της κοινότητας αυτής. Όπως γνωρίζουμε και όπως έχουμε ήδη δει σε πολλές μελέτες, οι νέοι που συμμετέχουν σε οργανώσεις νεολαίας έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να συμμετάσχουν και σε εκλογές στη συνέχεια και γενικότερα να συμμετάσχουν στα κοινά. Το καλό είναι πέρα από του νέου που συμμετέχουν. Είναι, είναι μάλλον ότι αυξάνεται ο αριθμό των νέων που συμμετέχουν. Η στρατηγική λοιπόν τη Ευρωπαϊκή Ένωση, από ό,τι φαίνεται, ήδη φέρνει κάποια αποτελέσματα σε κάποιε πτυχέ τη τουλάχιστον. Όμω θεωρώ ότι μπορούμε ε, βεβαίω να πάμε παραπέρα, μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερο αντίκτυπο, εάν μπορέσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να, να, να δούμε πώ θα συντονίσουμε τι πολιτικέ μα έτσι ώστε να έχουμε έναν αντίκτυπο πλέον συστημικό. Διότι η στρατηγική αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται κυρίω σε ένα πρόγραμμα, το, την εθελοντική υπηρεσία. Αυτό αφορά νέου, ε, λίγου νέου. Ο εθελοντισμό είναι κάτι το οποίο μπορεί να, με το οποίο μπορεί να ασχοληθεί ένα νέο στον ελεύθερο χρόνο του, στην τοπική του κοινότητα, ε, καθημερινά ή εβδομαδιαία. Ε, δυστυχώς η στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ήταν τα κατάλληλα για να, φτάσουν, να φτάσουμε ως όλους αυτούς τους νέους, ε, να τους προσεγγίσουμε και να τους δώσουμε μια ευρύτερη προοπτική. Με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, ε, αυτή τη στιγμή οι προχωρούν βέβαια, ελπίζω ε, με τη δική σας θέση να συνεισφέρετε και εσείς στην Επιτροπή Πολιτισμού για να πάμε ακόμα παραπέρα, να προχωρήσουμε και να προωθήσουμε την κινητικότητα και να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ένας πραγματικός συντονισμός των πολιτικών στην Ευρώπη, ώστε το κάθε κράτος μέλος να έχει ε, έναν νόμο ε, σε ό,τι αφορά τον εθελοντισμό, τους εθελοντές, και τα, δικαιώματά τους και να μπορεί ο κάθε νέος να, να συμμετάσχει σε μια τέτοια πρωτοβουλία. Τώρα, για τη δημοκρατική συμμετοχή των νέων. Ήταν ένα βασικό χαρακτηριστικό, ένα βασικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής, να εξασφαλίσει δηλαδή ότι οι νέοι θα συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ένα από τα βασικά αποτελέσματα, ένα από τα βασικά ζητήματα μάλλον είναι πώς θα έρθει κανείς σε επαφή με περισσότερους νέους, πώς θα φτάσει σε αυτούς. Και είναι σημαντικό αυτό όταν μιλάμε για δομημένο διάλογο, πώς θα μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτούς τους νέους. Χρειάζεται εδώ μια συστηματική προσέγγιση ε, συστηματική προσέγγιση στην δραστηριότητά μας. Είναι πολλοί οι νέοι οι οποίοι υποεκπροσωπούνται. Ε, πρέπει κανείς να ε, ενεργά να πάει στα σχολεία, να πάει στα κέντρα, να πάει στα, στα στρατόπεδα προσφύγων. δεν θα έρθουν από μόνοι τους όλοι αυτοί. Έχουμε πολλές πλατφόρμες επιγραμμικές, πολλά εργαλεία και μέσα με μια σειρά από hashtag, ε, τα οποία δυστυχώς δεν είναι και τόσο αποτελεσματικά για να έχουμε πρόσβαση σε αυτούς τους νέους. Πρέπει να πάμε πέρα από αυτήν την αυταπάτη ότι όλοι έχουν πρόσβαση στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Και εκεί αυτές οι οργανώσεις έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτούς τους νέους εκεί που ζουν, στην δική τους κοινότητα, στο δικό τους περιβάλλον. Υπάρχει το θέμα της ε, ανάπτυξης των τοπικών και εθνικών ε, συμβουλίων νεότητας ε, νεολαίας μάλλον, είναι σημαντικό να υπάρχει μια διαδικασία συμμετοχή, υπάρχουσα ε, διαδικασία σε περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαφορέ από χώρα σε χώρα σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Σε κάποιε χώρε ήδη ε, έχουν θεσπιστεί συμβούλια νεολαία ε, που συμμετέχουν συστηματικά στι διαβουλεύσεις για οποιαδήποτε νομοθεσία επηρεάζει τους νέους, αλλά σε κάποιες άλλες χώρες δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Θεωρούμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική πρέπει να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχει μια πραγματική διαδικασία παρακολούθηση σε συντονισμό με τα κράτη-μέλη για να εξασφαλίσουμε ότι αυτό θα γίνεται πιο συστηματικά. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει επίση μια πολύ καλή νομική βάση για να εξασφαλίσουμε μια πραγματική συμμετοχή με το άρθρο 165.2 τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Αυτό το άρθρο δίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δικαίωμα να εξασφαλίσει τη συμμετοχή των νέων στις δημοκρατικές διαδικασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή ο δομημένος διάλογος είναι το μόνο εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας. Δυστυχώς δεν αντιμετωπίζει όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το Εράσμους, την ε, πρωτοβουλία για την επασχόληση των νέων. Για όλα αυτά δεν προβλέπεται συμμετοχή των νέων. Είναι λοιπόν σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να πιέσει τα κράτη-μέλη να υπάρξει διαβούλευση με τους νέους για τις αποφάσεις που τους αφορούν, αλλά και να εξασφαλίσει συμμετοχή των νέων και στα δικά της προγράμματα τα ευρωπαϊκά. Με το δομημένο διάλογο είδαμε ότι είναι περιορισμένος ο χώρος που υπάρχει για μια πραγματική ευρωπαϊκή διάσταση. Ε, είναι λίγος ο χώρος που έχουμε εμείς, οι πρόσκοποι, δεν υπάρχει συστηματικό διάλογο ε, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σίγουρα λοιπόν υπάρχει περιθώριο βελτίωση. Ο δομημένο διάλογο ήταν ένα πολύ καλό εργαλείο έτσι ώστε οι νέοι να δικτυωθούν με τα Υπουργεία και τι γραμματείες νεότητα, νεολαία. Ε, χρήσιμο αυτό, διότι ορισμένε φορέ ο διάλογο αυτό δεν υπάρχει, αλλά πρέπει να πάμε ακόμα παραπέρα. Και τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στο ρόλο των οργανώσεων νεολαία στην εφαρμογή αυτή τη στρατηγική. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το ψήφισμά του 27 Οκτωβρίου 2016 σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της στρατηγικής ε, για την νεολαία ανέφερε ότι 57 οργανώσεις ε, θεωρούν ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία των νέων και, και ο λόγος τους κατά την θέσπιση νέων πολιτικών. Δηλαδή οι οργανώσεις των νεολαίων μας λένε ότι δεν συμμετέχουν επαρκώς στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ενώ εκπροσωπούν εκατομμύρια νέους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι στις οργανώσεις μας ε, ακολουθούμε δημοκρατικές διαδικασίες. Εξασφαλίζουμε ότι υπάρχει διαβούλευση των νέων τακτικά. Δυστυχώς από ό,τι φαίνεται συχνά η αξιοπιστία μας ως εκπρόσωποι των νέων ε, αμφισβητείται. Και αυτό είναι κρίμα, διότι εμείς εξασφαλίζουμε ότι λαμβάνουμε υπόψη μας ε, τις ανησυχίες των νέων, τα ζητήματα των νέων και προσπαθούμε να τις ε, μετατρέψουμε, να τις μεταφράσουμε σε συγκεκριμένες συστάσεις και σε συγκεκριμένες πολιτικές. Θέλει χρόνο για να μπορέσουν αυτές οι διαδικασίες να προχωρήσουν. Στις οργανώσεις νεολαίας εμείς ε, έχουμε μια προσέγγιση ε, μεταξύ ομοτήμων, μια εκπαίδευση, μια αγωγή αν θέλετε πολιτών με πολύ μικρό κόστος πολύ μικρό κοινωνικό κόστος και οικονομικό. Ταυτόχρονα βεβαίως πρέπει να μας να αναγνωριστούμε, να μας αναγνωρίσουν δηλαδή, να γνωριστεί αυτός ο ρόλος μας. Το 2018 ε, που είναι το έτος ε, για την ε, επικύρωση των άπτυπων δεξιοτήτων, ελπίζουμε να προχωρήσουμε, αλλά έως τώρα δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλο, μεγάλη ζέση για την επικύρωση, την αναγνώριση όλων αυτών των δεξιότητων που προκύπτουν από τέτοιου είδους ε, δραστηριότητε. Παρότι πρόκειται για κάτι που αποτελεί μέρο τη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να είναι προτεραιότητα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι πρόσφατε πρωτοβουλίε εκπαίδευση δεν αντιμετωπίζονται καθόλου. Δεν αντιμετωπίζουν καθόλου το θέμα του θελοντισμού. Δεν αναφέρεται καθόλου ε, το θέμα της άτυπης εκπαίδευση αναγνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει ανάγκη να επενδύσουμε ε, στην ε, εκπαίδευση των πολιτών, ε, ο ρόλος της άτυπης εκπαίδευσης, ο ρόλος των οργανώσεων νεολαίας δεν αναγνωρίζεται επαρκώς. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα κράτη-μέλη θα επενδύουν όχι μόνο στην τυπική εκπαίδευση, αλλά και στην άτυπη εκπαίδευση και στις οργανώσεις νεολαίας. Σε κάποιες χώρες πραγματικά είναι πολύ μικρή επένδυση στις οργανώσεις νεολαίας και αυτό τελικά οδηγεί στο ότι πολλές οργανώσεις νεολαίας ε, ε, χρησιμοποιούν ουσιαστικά το πρόγραμμα εράσμους ως βασικό εργαλείο, ως βασική πηγή χρηματοδότησης και οπότε τα προγράμματα αυτά πιέζονται οικονομικά. Θα πρέπει να υπάρξει μια σωστή, ένα σωστό εργαλείο παρακολούθησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να εξασφαλίσουμε ότι θα επενδύουμε πραγματικά ε, στην συμμετοχή των νέων διότι είναι αλήθεια ότι είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο, αλλά χρειάζεται στήριξη για να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση σε περισσότερους νέους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για την εισαγωγή που μας κάνατε και θα δοκιμάσουμε την διαδικασία. Και θα ήθελα να δώσω καταρχήν το λόγο στην εισηγήτριά μας και το Σκιώδης, αλλά όπως σας είπα θα το κάνουμε σε στυλ ping-pong, ερωταπαντήσεων δηλαδή, και της ενδότητας μια δεύτερη ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω λοιπόν και να θέσω ερωτήσει. Ε, συμφωνώ με αυτά που έλεγε η κυρία Ποτάρ για την ανάγκη να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή των ε, ε, οργανώσεων της νεολαίας και μεγαλύτερη εμπλοκή τους. Αλλά υπάρχει μία ε, πλευρά της κοινωνίας αυτών των νέων ανθρώπων που δεν ανήκει σε αυτές τις οργανώσεις των νέων, δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο α, αίτημα, γιατί μπορεί να έχει σπίτι και δουλειά, να μην έχει δηλαδή συγκεκριμένα αιτήματα ώστε να στρέφεται πιο συγκεκριμένα στα θεσμικά όργανα. Πώς μπορούμε λοιπόν να προσεγγίσουμε όλους αυτούς τους νέους που έχουν μια ζωή λίγο πολύ τακτοποιημένη και δεν νιώθουν την ανάγκη να ζουν σε μια κοινωνία και να συμμετέχουν σε προγράμματα εθελοντισμού. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο σκέλος των νέων που δεν συμμετέχει σε αυτά τα δίκτυα που έχουμε, ούτε από θεσμική σκοπιά και ούτε ε, σε οργανώσεις ε, της νεολαίας. Πώς μπορούμε λοιπόν να εμπλέξουμε και αυτό το σκέλος τη κοινωνία. Θαυμάσια. Παρακαλώ, κυρία Ποτάρ. Παρακαλώ, κυρία Ποτάρ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι αυτή είναι πολύ ευστοχή ερώτηση. Καταρχάς, ε, να πω ότι ελπίζουμε να υπάρξει μεγαλύτερη δέσμευση των νέων ε, σε οργανώσεις νεολαίας, όχι μόνο των νέων απαραίτητα, μπορεί να συμμετέχουν στον αθλητισμό, σε άλλες εθελοντικέ οργανώσει. Και πιστεύω ότι η κοινωνία εν γέννη ε, θα πρέπει να θεωρεί αυτή τη δέσμευση κάτι πολύτιμο. Ε, δεν είναι οι οργανώσει των νέων μόνο αυτές οι οποίες ε, διαδραματίζουν κομβικό ρόλο. Ε, συμφωνώ μαζί σα ότι έχουν κάθε δικαίωμα οι νέοι άνθρωποι να μην συμμετέχουν και να μην κάνουν τίποτα. Αλλά πιστεύω ότι τα τοπικά συμβούλια νεολαία και τοπικά φεστιβάλ νεολαία μπορεί να είναι χώρες στου οποίου οι νέοι ε, μπορεί να ε, έχουν λόγο και να ακουστεί η φωνή τους και ε, χώρες στους οποίους οι νέοι εκφράζουν τις απόψεις τους. Έχουμε δει σε διαδικτυακές έρευνες αντίστοιχες απαντήσεις. Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι λοιπόν να εισακουστεί η άποψή τους. Αλλά εμείς από πλευρά μας θεωρούμε ότι η δέσμευση της νεολαίας ε, με οποιαδήποτε μορφή είναι κάτι θετικό ε, και πρέπει να πάμε πέραν του να ακούμε απλώ τι έχουν να μας πούνε, να συμβάλλουν και με θετικό τρόπο στην κοινωνία. Ευχαριστώ. Άλλες ερωτήσεις. Εντάξει. Προχωράμε λοιπόν. Με τον κύριο Μάλινοφ. Καταρχήν οι συγητές εισηγητέ και σκιώδεις. Κύριε Μάλινοφ, θέλετε να πάρετε το λόγο. Τότε η κυρία Μίχελς έχει το λόγο. Ούτε εσείς. Η Χέλγα Τρούπελ δεν είναι εδώ. Τότε θα συνεχίσουμε με τη Σίλβια Κώστα. Ε, Χάρηκα που άκουσα την παρουσίασή σας. Γνωρίζω πολύ καλά το κίνημα των προσκόπων και το παρακολουθώ εδώ και χρόνια. Μία ερώτηση προτεραιότητε για τη νέα στρατηγική για την νεολαία. Όπω γνωρίζετε έχουμε μια εξαιρετική συγκήτρια και θέλουμε να έχουμε μια πολύ καλή έκθεση τη Επιτροπή που να αποτελέσει και όθηση. Κάποια πράγματα τα είπατε, συμμετοχή στην κοινωνία κλπ. Ποια είναι η, η άποψή σα για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύη και το σχετικό πρόγραμμα. Εμεί έχουμε διάθεση να ε, λάβουμε υπόψη μας τα στοιχεία του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης σε τρίτες χώρες και να υπάρχει και μεγάλη συμμετοχή στα δίκτυα ε, των ενώσεων της νεολαίας ως ε, στοιχείο εμπειρογνωμοσύνης. Ε, τι θεωρείτε ότι μπορεί να προσφέρει περισσότερο το Ευρωπαϊκό Σέμα Αλληλεγγύης, το οποίο εμείς θα αποκαλέσουμε η υπηρεσία σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντισμού. Ευχαριστώ. Πολύ καλή ερώτηση. Όπως ανέφερα, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα περιλαμβάνει αυτό που αποκαλούσαμε την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία. Και είναι πολύ καλό εργαλείο. Ε, αλλά πέραν αυτού πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε τον εθελοντισμό ως ε, ε, στρατηγική πολιτική. Υπάρχει ήδη ανοιχτός μέθοδο, ανοιχτή μέθοδος συντονισμού στην παιδεία, αλλά δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στον εθελοντισμό. Και πιστεύω ότι αυτό το σώμα αλληλεγγύης θα πρέπει να περιλαμβάνει αυτή την πτυχή και να εξασφαλίσουμε και ότι οι διεθνείς και εθνικές οργανώσεις που έχουν και διάσταση εθελοντισμού θα μπορούν να συντονιστούν ε, και να χρησιμοποιήσουν νέα εργαλεία για τη διαχείριση του εθελοντισμού και ε, να προσπαθήσουμε να δούμε την ε, πολιτική εθελοντισμού και νομοθεσία για τον εθελοντισμό. Αυτά πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και νομίζω ότι αυτό αποτελεί και ευκαιρία να πάμε πέραν της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας. Σίλβια, έχεις κάποια ερώτηση επιπλέον? Να ρωτήσω μόνο εάν για σας ε, ο εθελοντισμός θα πρέπει να είναι αυτό που προέχει ή να είναι η πλήρης ε, ε, πτυχή της αλληλεγγύης. Ξέρετε ότι εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να προέχει ο εθελοντισμός και όχι η εργασία. Θεωρώ ότι είναι πολύ πολύτιμο να υπάρχει αυτό το εργαλείο γιατί είναι ένα στοιχείο κινητικότητας που μπορούν να, αντιμετωπίσουν, να χρησιμοποιήσουν και χώρες ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω όμως ότι το μισό τουλάχιστον πρόγραμμα θα πρέπει να έχει ε, μια ευρύτερη διάσταση. Ίσως το μισό να είναι ε, θελοντισμός και το άλλο μισό να είναι συντονισμός, πολιτική, να φροντίσουμε όντως ότι θα είναι ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα. Ευχαριστούμε. Ε, Μιχαέλα. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτά τα εισαγωγικά λόγια. Συγγνώμη που καθυστέρησα λίγο. Αλλά θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Νεότητας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Και μάλιστα σε συνεργασία με εσά, δηλαδή με ευρωπαϊκές οργανώσεις της ε, νεολαίας. Ε, λέτε τι λέψεις εντοπίζετε κλπ. Και ε, αυτό είναι σημαντικό και εσά να διαβάσετε ε, τις πληροφορίες αυτές, δηλαδή ότι υφίσταται αυτή η στρατηγική και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να προσφέρει κάτι στους νέους. Τώρα, όσον αφορά τη χρηματοδότηση, πιστεύω ότι οι νέοι άνθρωποι είναι εκείνοι που μπορούν, είναι σε θέση από ένα ευρώ να κάνουν δέκα ευρώ. Και θα ήθελα να τονίσω ότι εδώ πρόκειται για μια επένδυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, νεολαία της Ευρώπης που είναι σε θέση να πολλαπλασιάσουν το κάθε ευρώ και να το εξοπλίσουν. Τώρα, ως προς το ερώτημα τι να κάνουμε για τους νέους που δεν είναι οργανωμένοι οι άλλοι που είναι οργανωμένοι είτε σε προσκοπικές οργανώσεις είτε σε άλλες, αυτοί μπορούν να συνεργαστούν και είναι σε θέση να προσφέρουν συνεργασία φιλία σε νέους που μέχρι τώρα δεν την έχουν βρει. βρει. Ο κάθε νέος άνθρωπος χρειάζεται φίλους, συντρόφους κλπ. Άρα λοιπόν οι οργανώσεις αυτές μπορούν να ωφελήσουν νέους που δεν έχουν ριζώσει πουθενά αλλού. Um, Πιστεύω ότι σε τοπικό επίπεδο μπορούμε να έχουμε κέντρο νεότητας και ε, εργαζόμενους με τη νεότητα ε, στο επίπεδο της ε, κοινότητας πέρα από τις οργανώσεις των νέων. Και όπως είπαμε προηγουμένως, ε, μπορούν να διοργανωθούν φεστιβάλ νέων κλπ. όπου οι νέοι μπορούν ε, να εισακωστούν και να έχουν όλες τις δυνατότητες. Αλλά πέρα από αυτό, οι, νεότητες, οι οργανώσεις νεότητας χρειάζονται μια υποστήριξη. Γιατί δεν έχουν πολλές δυνατότητες να συστήσουν νέες ομάδες, να δημιουργήσουν νέες δομές σε κοινότητες εκεί όπου δεν υφίστανται ήδη. Ευχαριστούμε πολύ. Αφού δεν ε, υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις, έχω εγώ μία ερώτηση για το διαρθωμένο διάλογο. Ε, ποια είναι η δική σας εμπειρία με τον διαρθωμένο διάλογο την περασμένη χρονιά. Γιατί θυμάμαι ότι στην αρχή όταν ξεκινήσαμε να το συζητούμε υπήρχε μεγάλη ανησυχία ότι αυτή η προσέγγιση δηλαδή ενδιαφερόμενους διάλογο από τοπικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό το οποίο συζητείται σε ε, τοπικό επίπεδο δεν έφτανε ποτέ στο επίπεδο της ε, Ένωσης και κάπου χανόταν ενδιάμεσα. Ποια είναι η δική σας εμπειρία? Um, Καταρχήν, νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον να συζητήσουμε το θέμα αυτό, γιατί υποτίθεται ότι θα πρέπει να συζητούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τοπικά θέματα. Το τοπικό συμβούλιο και οι τοπικές πλατφόρμες βεβαίως θα ήταν πιο ενδεδειγμένες για να συζητήσουν τοπικά θέματα. Και θα πρέπει βεβαίως να εξασφαλίσουμε και το ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά είναι πιο σημαντικό σε κάθε επίπεδο να δημιουργείται μια προστιθέμενη αξία. Πιστεύω ότι ο διαφρομένος ε, διάλογος είναι σημαντικός και όλοι προσπαθούμε να έχουμε διαβιλεύσεις σε όλα τα επίπεδα, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι ότι ε, συμμορφωνόμαστε με τις προοπτικές της, ε, πολιτικής για τους νέους. Ε, δεν ξέρω, το θέμα είναι κατά πόσο είναι αποτελεσματικό να συζητήσουμε ένα θέμα σε όλα τα επίπεδα. Ίσως ε, δεν είναι δυνατόν. Το μία ερώτηση. Ποια θα ήταν η... η ορθή προσέγγιση για το διορθωμένο διαρθρωμένο διάλογο. Θα ήταν σωστό να υπάρχει κάθε χρόνο ένα συγκεκριμένο θέμα αντί να λέμε ότι το, ο διαρθρωμένος διάλογος θα πρέπει κάθε φορά να αποφασίζει για ποιο θέμα θεωρούν σημαντικό. Ίσως θα έπρεπε το ευρωπαϊκό επίπεδο να διατυπώνει ποιο είναι το σημαντικό θέμα για το διαρθρωμένο διάλογο και στα άλλα επίπεδα. Το θεωρείτε σωστό. Ακούστε, ήταν ενδιαφέρον να επικεντρωθούμε, να εστιάσουμε εκεί που πρέπει, διότι δάλος ε, οι συστάσεις δεν θα ήταν αρκετά συγκεκριμένες. Βεβαίως, εξτάσαμε το θέμα της σημασίας του επίπεδου, αλλά επειδή οι ήταν πάντα καλές, η ανησυχία μας ήταν η εφαρμογή. Και εφαρμογή δυστυχώς είχαμε λίγη, καθώς και παρακολούθηση δεν είχαμε επαρκή για το τι γίνεται τελικά στην πράξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο δομημένος διάλογος λοιπόν είναι κατά κάποιο τρόπο μία συνάντηση όπου συζητούμε κάποια πράγματα αλλά δεν, είναι πραγματι... δεν σημαίνει πραγματική συμμετοχή των νέων. Ευχαριστούμε. Νομίζω ότι λειτουργήσε καλά το πράγμα για αυτό το πρώτο γύρο. Και τώρα θα περάσουμε στο δεύτερο προσκεκλημένο μας, τον κύριο Μαγιάμα, ε, μέλος του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τους Νέους. Και εσείς έχετε το λόγο για 10 λεπτά κι εσείς. Hello everyone. Καλημέρα σε όλους. Το όνομα μου είναι Βίλε Μαγιάμα. Προσπαθώ να κάνω παρουσιαστώ, προέρχομαι από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νέων, είμαι και εθελοντής, είμαι και νέος. Ε, για όσους δεν γνωρίζουν το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νέων, είμαστε μια πλατφόρμα όπου συμμετέχουν πάνω από 100 οργανώσεις νέων, ε, συμβούλια ε, και διεθνείς οργανώσεις. Για το θέμα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής ξεκινήσαμε ε, το 2016 το θέμα τη Ευρωπαϊκή Στρατηγικής Νέων και ό,τι σα πω τώρα αποτυπώνει τι συζητήσει που είχαμε με τι οργανώσει μέλη μα που εκπροσωπούν του νέου ανά την Ευρώπη. Ε, πιο συγκεκριμένα σήμερα εξετάζουμε τη διατομεακή προσέγγιση, την σφαιρική προσέγγιση, για την πολιτική νεολαία και ελπίζουμε να είναι χρήσιμη για εσά. Λοιπόν, τι σκόπευα να πω σήμερα. Θα ξεκινήσω με το τι εννοούμε όταν λέμε πολυτομιακή πολιτική. Στη συνέχεια θα σας πω πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, τι μένει να βελτιωθεί και στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε κάποιες ιδέες για το τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα και τέλος να μην ξεχανάμε ότι ο στόχος ε, η πολιτομιακή πολιτική δεν είναι αυτό ο σκοπός, είναι ένα εργαλείο έτσι ώστε να πετύχουμε του ευρύτερου στόχου μα. Πρόκειται για μια μικρή υπενθύμηση, λέει, στο τέλο ε, του νόήματο του ολοχηρήματο. Λοιπόν, τι εννοούμε όταν λέμε πολυτομιακή. Όταν μιλάμε για πολιτομιακή πολιτική νέων, σημαίνει ότι χρειάζεται ένα κατάλληλο συντονισμό μεταξύ των διαφόρων δημοσίων φορέων που είναι υπεύθυνοι ε, για ζητήματα που αφορούν του νέου. Οι διάφορε δημόσιε αρχέ που ασχολούνται με ζητήματα που επηρεάζουν τους νέους πρέπει να εργαστούν από κοινού για την θέσπιση και την παρακολούθηση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση αυτών των πολιτικών. Υπάρχει μια αναφορά ε, στα οχτώ πρότυπα ε, για το πώς ορίζεται η ποιοτική πολιτική νεολαία, νεολαίας και μια, ένα από τα τρία αυτά είναι η πολιτομιακή προσέγγιση. Εκεί αναφερόμαστε σε τρεις δείκτες για να μπορέσουμε να μετρήσουμε κατά πόσο όντω λαμβάνει η χώρα διατομιακή ε, πολιτική ποιότητα. Πρέπει να υπάρχει καταρχήν συνεργασία μεταξύ όλων των τομέων. Θα επανέλθω για το τι σημαίνει αυτό. Δεύτερον, θα πρέπει τα ζητήματα των νέων να διέπουν όλους τους τομεί πολιτικής. Και τρίτον, η αξιολόγηση της πολιτικής νέων να χρησιμοποιείται για να μαθαίνουμε μεταξύ ομοντήμων ε, στους διάφορους τομείς. Αυτό εννοούμε όταν λέμε διατομιακή. Τι συμβαίνει λοιπόν αυτή τη στιγμή. Η στρατηγική νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει την ανάγκη πολυτομιακών προσεγγίσεων και του mainstreaming των νέων ε, και η παρακολούθηση της εφαρμογής από τα κράτη-μέλη. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή έχουμε πετύχει το στόχο μας. Η στρατηγική επίσης αναφε... έχει, και μια οριζόντια προσέγγιση και, και οριζόντια προσέγγιση και κάτι προσέγγιση για να παίξει ένα mainstreaming των ζητημάτων νεολαίας σε διάφορους τομείς. Σε οριζόντιο επίπεδο έχουμε την εκπαίδευση, την απασχόληση, την υγεία κτλ. Σε κάθε το επίπεδο ε, έχουμε τα ζητήματα ε, που εστιάζουν στους νέους, δημοκρατική συμμετοχή ή εθελοντισμός. Πέρα από αυτόν, αυτή την, πολιτικό στόχο, η αξιολόγηση της στρατικής νεολαίας, την οποία αναφέρθηκαμε προηγουμένως το 2016, δείχνει ότι πιο πολύ είχε αντίκτυπο το ξεκάθετο επίπεδο και όχι στο οριζόντιο επίπεδο. Υπάρχουν δηλαδή κάποια θετικά μηνύματα, αλλά μένει ακόμα πολλή δουλειά. Μια σειρά από χώρε ε, στην ίδια έκθεση ε, αναφέρουν ότι έχει βοηθήσει η στρατηγική αυτή σε μια καλύτερη πολυτεμιακή συνεργασία. Μπορώ να δώσω και παραδείγματα σχετικά τα οποία θα μπορούσαν να χρήσουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σχετική συζήτηση. Οι πιο κοινέ δράσει, οι πιο συνηθισμένε ε, είναι η δημιουργία κάποιων πολυτομιακών ε, δομών μεταξύ διαφορών υπουργείων. Ε, στη Σουηδία, παραδείγματος χάρη, στην νομοθεσία υπάρχει ένας ε, νόμος που επικεντρώνεται στην, στους νέους, στην, στις, σωστές, στις σωστές συνθήκες εργασίας. Αναφέρει ρητά δηλαδή ο νόμος ότι η πολιτική νεολαία είναι διατομιακή και αναφέρει μάλιστα νομοθεσία ποιοι είναι οι τομεί που πρέπει να αφορά. Εκπαίδευση, απασχόληση, στέγαση, υγεία, πολιτισμός και ψυχαγωγία. Να ένα παράδειγμα από το Βορρά λοιπόν. Ε, υπάρχουν κάποιες εξελίξεις, ε, υπάρχουν κάποιες καλές πρακτικές, όμως η, η σφαιρική εικόνα είναι αρκετά άνηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, σε θεσμικό ευρωπαϊκό επίπεδο, ήδη στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2009 για την στρατηγική νεολαία της Ένωσης, η διατομιακή προσέγγιση αναφέρεται ρητά τέσσερις φορές. Το mainstreaming των νέων αναφέρεται πέντε φορές. Δεν είναι θέμα να το λέμε λοιπόν σε ένα κείμενο ή να συμφωνούμε επί της αρχής ότι είναι σημαντικό. Είναι θέμα το να βρεθούν τα κατάλληλα εργαλεία ή να βελτιωθούν τα υπάρχοντα εργαλεία έτσι ώστε αυτή η φιλοδοξία την οποία έχουμε εκφράσει να πάρει σάρκα και οστά. Πώς θα το κάνουμε λοιπόν αυτό. Εδώ έχουμε τις απαντήσεις. Τώρα, με βάση τις συζητήσεις που είχαμε με τα μέλη μας, ε, προκύπτουν τα εξής, χαίρομαι ιδιαίτερα που τα μοιράζομαι μαζί σας και είμαι, θα ήμουν ευτυχής να τα συζητήσουμε και όλες. Καταρχήν να εφαρμόσουμε τα youth checks. Εσείς να εφαρμόσετε τα youth checks, δηλαδή. Ε, μέσω αξιολόγησης ε, αντικτύπου για τους νέους και μέσω της εφαρμογής της νομοθεσίας. Η Αυστρία, παραδείγματος χάρη, το κάνει ήδη αυτό. Είναι μια πρακτική που λαμβάνει η χώρα σε κάποια κράτη-μέλη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίση ω θεσμικό όργανο θα μπορούσε να είναι ένα από τα όργανα που θα αξιολογεί τον αντίκτυπο τη κάθε πρόταση που προέρχεται από το ευρωπαϊκό επίπεδο και που επηρεάζει του νέου. Ένα άλλο σημείο. Ε, θα πρέπει να έχουμε την ίδια προσέγγιση με τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά το, διαθεσμι... το διαθεσμικό συντονισμό και τη δημιουργία σχετικών οργάνων. Να γίνει αυτό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να εμπνευστούμε από τα κράτη-μέλη, να δημιουργηθεί μια διαθεσμική ε, ομάδα εργασίας ε, όπου θα συμμετέχουν τα κράτη-μέλη, η Κομισιόν, η Επιτροπή των Περιφερειών, η ΕΟΚΕ, το Κοινοβούλιο και κυρίως βέβαια οι εμπλεκόμενοι φορείς αυτών των πολιτικών, οι ίδιοι οι νέοι οργανώσεις νέων αυτές καθ' αυτές. Μια τέτοια ομάδα θα μπορούσε να ε, βοηθήσει στον να καλύτερο συντονισμό, καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών. Τρίτον, το τριετές πρόγραμμα εργασιών που ήδη αποτελεί μέρος ε, της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Νέων θα πρέπει στο μέλλον ε, να αποσαφινιστεί. Να ξέρουμε δηλαδή ποιοι συμμετέχουν και ποιες είναι οι ευθύνες τους. Αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ήδη στο σχέδιο το τριετές. Και κάτι που προκύπτει από την αξιολόγηση είναι η σύσταση να συνεχιστεί το mainstreaming των νέων σε άλλους τομείς πολιτικής. Δεν μιλάμε εδώ για ένα κατάλογο νέων τομέων, αλλά να αναπτύξουμε συγκεκριμένους στόχους πολιτικής στους συγκεκριμένους τομείς. Η ποιοτική πολιτική για τους νέους ε, θα πρέπει να οδηγήσει σε στόχους οι οποίοι είναι μετρήσιμοι, οι οποίοι επίσης να κοστολογούνται σε οριζόντιο επίπεδο θα πρέπει να συμπεριληφθούν εδώ βεβαίως και οι βασικοί δικαιούχοι, ε, οι νέοι, δηλαδή να συμμετέχουν στην θέσπιση των στόχων αυτών. Τώρα, η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού μας δίνει κάποια παραδείγματα. Εμείς θεωρούμε ότι τα εθνικά σχέδια δράσης, τα οποία ήδη αποτελούν μέρος μιας ανοιχτής μεθόδου συντονισμού, όχι στον τομέα της νεολαίας βέβαια, θα μπορούσαν να εισαχθούν και στον τομέα της νεολαία και των νέων. Ε, πράξη τα εθνικά σχέδια δράση ε, θεσπίζονται από τα κράτη-μέλη και αναφέρουν πώ τα κράτη-μέλη θα πετύχουν του στόχου που αναφέρονται στη στρατηγική για του νέου. Αυτό θα βοηθήσει την παρακολούθηση τη διαδικασία αλλά και τη διασύνδεση μεταξύ των διαφόρων φορέων σε διάφορα επίπεδα, να υπάρχει δηλαδή μια κάποια συνοχή όταν μιλάμε για την πολιτική για του νέου στην Ευρώπη. Οι οργανώσει νέων θα πρέπει βεβαίω να συμμετέχουν στην θέσπιση αυτών των σχεδίων δράση. Έχω ακόμα ένα λεπτό. Ε, το να βάλουμε τους νέους ε, στην καρδιά ε, των πολιτικών που τους αφορούν δεν είναι απλά μια ωραία ιδέα. Έχει και αντίκτυπο ε, πραγματικό. Γνωρίζουμε ότι οι νέοι έχουν δικαιώματα, το λέμε, αλλά στην πράξη πολλοί νέοι αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλη δυσκολία στον έχουν πρόσβαση στα δικαιώματα αυτά. Ε, έχουμε κάποια στατιστικά στοιχεία τα οποία είναι απαράδεκτα. Πρέπει σίγουρα να κάνουμε περισσότερα και κάποια από τα εργαλεία που, υπάρχουν, που έχουμε στη διάθεσή μας δεν λειτουργούν. Βεβαίως, ε, τουλάχιστον υπάρχει η πολιτική φιλοδοξία για το mainstreaming, για τη διατομιακή προσέγγιση. Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνουν αυτά. Τώρα η νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική Νέων είναι μια ευκαιρία έτσι ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει αυτέ και να δείξουμε ε, στου ε, νέου Ευρωπαίου ότι η Ευρώπη νοιάζεται για αυτού, του προσφέρει ευκαιρίε, του ακούει και τους ε, δέχεται να συμμετέχουν στη διαδικασία. Σας ευχαριστώ πολύ. vielen Ευχαριστούμε πολύ. Και θα ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία όπως προηγουμένως. Το λόγο έχει η συγγέτριά μας. Ναι, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Με το Youth Forum είναι αλήθεια ότι πολλές φορές συζητήσαμε την πολιτική της νεολαίας και πράγματι τουλάχιστον ε, στη συζήτηση έχουμε κερδίσει και όλοι αντιλαμβάνονται ότι η πολιτική για την νεολαία πρέπει να είναι ε, προτεραιότητα και να είναι και εγκάρσια προτεραιότητα. Ε, αλλά ακόμα δεν έχουμε βρει τα κατάλληλα μέσα για να το υλοποιήσουμε στην πραγματικότητα. Είναι η ίδια συζήτηση που γίνεται με τις πολιτικές του φίλου. Ναι, μεν έχουμε κερδίσει στα λόγια, αλλά ακόμα δεν έχουμε βρει τον τρόπο να το υλοποιήσουμε στην πράξη. Ε, από τις προτάσεις ε, για την νεολαία που ε, αφορά και το Youth Check που γίνεται ήδη στην Αυστρία. Ε, θα πρέπει λίγο να συζητήσουμε τα κριτήρια και τους δείκτες που χρησιμοποιούνται για, αυτούς, για αυτά τα Youth Checks για να δούμε πώς γίνονται αυτές οι πολιτικές ε, και αν γίνονται πραγματικά πολιτικές οι οποίες είναι οριζόντιες. Και το ίδιο αφορά και τους πιο συγκεκριμένους στόχους. Υπάρχουν ήδη συγκεκριμένες ε, προτάσεις όταν αναφέρεστε σε συγκεκριμένους στόχους, ε, αναφέρεστε σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς που είναι εγκαταλελειμμένοι όσον αφορά την πολιτική της νεολαίας. Γιατί είναι αλήθεια ότι για την απασχόληση πάντα μιλάμε για την νεολαία, για τα ανθρώπινα δικαιώματα για την νεολαία, αλλά μπορεί να υπάρχει για παράδειγμα τομέα της υγείας ή κάποιων ελευθεριών που ε, θα μπορούσαμε να αναζητήσουμε κάποιους πιο συγκεκριμένους στόχους. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η απάντηση αυτή ενισχύει ακριβώς το γεγονός ότι ε, συμφωνούμε ως προς το που θέλουμε να πάμε, αλλά ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα φτάσουμε εκεί. Ε, όσον αφορά τα youth checks πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκα στην Αυστρία ως παράδειγμα, υπάρχουν και άλλα κράτη-μέλη όπου ήδη εφαρμόζεται αυτό ε, και αυτή η συζήτηση γίνεται με τα Εθνικά Συμβούλια Νεολαίας, τα οποία αναφέρθηκαν ήδη. Ε, και αυτό είναι κάτι το οποίο προκύπτει και από τα όσα μας ε, λέτε εδώ στην αίθουσα και φαίνεται ότι είναι θετικό και θα μπορούσαμε ίσως να το χρησιμοποιήσουμε και να δούμε πώς μπορούμε να το προσαρμόσουμε ε, στο πλαίσιο της νεολαίας. Δεν θα ήθελα να δοθεί εδώ η εντύπωση ότι η λύση αυτή είναι πανάκια για τα πάντα, ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε το αυστριακό σύστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τα μέλη από την Αυστρία έχουν ιδέες για το πώ ε, θα μπορούσε να εφαρμοστεί και με διαφορετικό τρόπο στην ίδια την Αυστρία. Η συζήτηση δηλαδή είναι σε εξέλιξη, αλλά ακόμα δεν έχουμε καταλήξει το συμπέρασμα για να πούμε ότι αυτό είναι το συγκεκριμένο σύστημα που πρέπει να προσαρμοστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά από τα όσα μου φαίνεται ότι λαμβάνω ως μήνυμα από εσά είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Τώρα, ε, ως προς το πού μπορούμε να πάμε για την πολιτική για την νεολαία. Πρόκειται για πάρα πολύ ευρύ τομέα. Και ο μόνος τρόπος ε, που θα μπορούσα να σκεφτώ είναι να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι ε, εν μέρη όσον αφορά το θέμα, δηλαδή ε, εξαρτάται το παράδειγμα βέβαια και από το επίπεδο το οποίο συζητάμε, το, σε τοπικό επίπεδο είναι διαφορετικές αρμοδιότητες, ε, αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν συμμετέχουμε ε, σε πολλές από τις συζητήσεις που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η νεολαία δηλαδή ως ένα ενδιαφερόμενο μέρος ε, με συμμετοχικό τρόπο συμμετέχει σε συζητήσεις για την παιδεία, για την εθελοντισμό, την ε, διαβίου μάθηση και τη συμμετοχή. Αλλά για παράδειγμα υπάρχουν συζητήσεις για το μέλλον της Ευρώπης, για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση κλπ που υπάρχει χώρος για άλλους, αλλά όχι και τόσο πολύ για μας. Αυτή λοιπόν είναι η πιο άμεση τομή στους οποίους ε, θα συμμετέχαμε με τα χαράς ε, και θεωρούμε ότι γενικότερα είναι οι άνθρωποι θα συμμετείχαν. Η κυρία Νηριάδα. Για ένα λεπτό. Ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση και μου αρέσει η ιδέα ότι υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση, γιατί αυτό συμπεριλαμβάνει τα πάντα, αλλά ταυτόχρονα θεωρώ ότι μια προσέγγιση η οποία βασίζεται στα δικαιώματα είναι καλή προσέγγιση, γιατί καλύπτει αυτή την ολιστική προσέγγιση. Και κάτι στο οποίο νομίζω θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε όλοι είναι το θέμα τη ψυχική υγεία σε ευρωπαϊκό τομέα διότι σε εκπαιδευτικό επίπεδο έχουμε διαφορετικού στόχους από χώρα σε χώρα, αλλά όσον αφορά την ψυχική υγεία, τα θέματα νομίζω ότι είναι ταυτόσιμα. Και εγώ ως Ιρλανδή Ευρωβουλευτή, θεωρώ ότι είναι ένα τεράστιο ζήτημα το γεγονός ότι έχουμε τόσο μεγάλο αριθμό αυτοκτονιών νέων ανθρώπων. Ε, και αυτό είναι κάτι το οποίο συζητούμε πολύ συχνά εδώ, πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε τους νέους ανθρώπους, να επενδύσουμε στους νέους και στην παιδεία τους, λες και είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ μακρινό, ε, ενώ το πρόβλημα είναι ε, εδώ και τώρα. Δεν είναι κάτι που αφορά το μέλλον, είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή. Ε, με ενδιαφέρουν τα youth checks και πώς θα μπορέσετε να έχετε κάποιο αντίκτυπο εδώ και όσον αφορά τα ε, συμβούλια νεολαίας στην Ιρλανδία νομίζω ότι υπάρχει έλλειμμα για την ίση πρόσβαση σε εκπαίδευση και επιβαρύνονται οι νέοι άνθρωποι με δάνεια πριν ακόμα ολοκληρώσουν τις σπουδέ τους. Είναι ήδη χρεωμένοι. Και μπορούν να γίνουν πολλά λοιπόν για την πολιτική. Ευχαριστώ για την παρέμβασή σας και με τα χαράς ε, να δω και κάποια πρόοδο, γιατί ξέρω ότι είναι και μια ε, πολιτική ενεξελίξη. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Έχω το αρχικό ψήφισμα της οργάνωσής μας από το 2016 Υπάρχει μια ολόκληρη ενότητα εδώ στο έγγραφο η οποία αναφέρεται στις αρχές ε, του γεγονότος ε, στι αρχέ συγγνώμη, στι οποίε θα πρέπει να εδράζεται η πολιτική μα, χωρί να επισέλθουμε σε λεπτομέρειε. Ε, ένα από τα βασικά πρότυπα τα οποία έχουμε καθορίσει είναι μια προσέγγιση βάσει δικαιωμάτων. Για μα αυτή είναι η σωστή λύση για να κάνουμε πολιτική. Αν πετάμε από κρίση σε κρίση, προσπαθώντα απλώ να σβήσουμε φωτιέ, κάπου θα πάμε, αλλά δεν θα είναι όμορφα. Ε, θέλουμε ένα πιο στρατηγικό τρόπο σκέψη και πιο βιώσιμο τρόπο σκέψη, και πρέπει λοιπόν να ε, θεμελιώσουμε τις πολιτικές μας και τα δικαιώματά μας. Και επ' αυτού συμφωνούμε. Όσον αφορά το σχόλιο για την ψυχική υγεία και την εκπαίδευση και τα δύο θέματα αυτά και όσον αφορά τις αρχές της ουσίας της πολιτικής περιλαμβάνονται στην αρχική μας πρόταση και θα ήταν ενδιαφέρον ίσως να συζητήσουμε λίγο πιο αναλυτικά πώς μπορούμε να καθορίσουμε και αυτούς τους στόχους. Όσον αφορά το θέμα των δανείων, και εγώ έχω φοιτητικό δάνειο, δεν έχω αποφοιτήσει και προσβλέπω ε, στην αποπληρωμή του με την πρώτη μου θέση εργασίας. Ευχαριστώ. Η μας, ε, ε, μας ε, χτυπάει όλους κάποια στιγμή, αλλά αυτό δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Θα έπρεπε η εκπαίδευση να είναι δωρεάν και προσβάσιμη για όλους. Ευχαριστώ πολύ. εκτιμώ την εργασία σας σαν μια ομπρέλα για, για το, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Φόρουμ της Νεολαίας θεωρώ ότι υπάρχει πολύ καλή συνεργασία και εκτιμώ την προσέγγισή σας γιατί είναι πολύ καλά δομημένη και συστηματική. Ποια είναι η γνώμη σας για την εγγύηση για την νεολαία ως πρόγραμμα. Ο στόχος αυτού του προγράμματος είναι να βοηθήσει την νεολαία να βρει απασχόληση. Θέση απασχόλησης. Ε, τώρα σκεφτόμαστε, προβληματιζόμαστε κατά πώς θα έπρεπε να αλλάξουμε αυτό το πρόγραμμα. Τι σύσταση θα μπορούσατε να μας κάνετε, γιατί θα ήταν χρήσιμο να μας δώσετε τη γνώμη σας. Παρακαλώ. Ναι, μου αρέσει αυτό το ερώτημα. Είχαμε μια συνάντηση αυτό το Σαββατοκύριακο και περάσαμε ώρες να συζητούμε την ε, εγγύηση για τους νέους και το μέλλον της. Ε, υπάρχει ένα έγγραφο επ' αυτού. Δεν έχω το χρόνο βεβαίως να σας το παρουσιάσω σημείο προς σημείο, αλλά ε, να αναφερθώ στα σημεία κλειδιά. Το πρώτο μάθημα είναι ότι πρόκειται για μια καλή πρωτοβουλία. Το πρώτο που πρέπει να πούμε, διότι έχουν ακουστεί πολλές κριτικές. Για μας όμως είναι μια αναγνώριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το θέμα της νεολαίας είναι ένα ζήτημα ε, όπου αξίζει να γίνουν επενδύσεις και η εγγύηση για τους νέους είναι ένα παράδειγμα προς την κατεύθυνση αυτή. Τώρα, για να φτάσουμε σε ένα πιο ρεαλιστικό επίπεδο, η εφαρμογή είναι εξαιρετικά άνηση, διότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε να δώσουμε μια κατεύθυνση για τη χρηματοδότηση. Αλλά το τι γίνεται μετά εξαρτάται από το εθνικό επίπεδο και εκεί μένουν πάρα πολλά να γίνουν. Ε, δεν μπορώ βεβαίως να σας δώσω κάποια μαγική λύση για το πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί καλύτερα. Ε, επίσης να πω ότι βεβαίως εκτιμούμε την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και την σημασία που δίνεται στους νέους. Το θέμα της ανεργίας των νέων δεν μπορεί να συζητηθεί ή να λυθεί μάλλον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειάζεται επένδυση σε εθνικό επίπεδο, χρειάζεται δέσμευση σε εθνικό επίπεδο. Δεν πρέπει να προσπαθήσουμε να παίξουμε το ρόλο αυτό εμείς. Στα κράτη-μέλη ε, εναπόκειται ο ρόλος αυτός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθήσει, να καλύψει τα κενά Ταυτόχρονα όμως πρέπει να ζητήσουμε περισσότερες επενδύσεις για τους νέους σε εθνικό επίπεδο. Να το ζητήσουμε περισσότερο από ό,τι το πράττουμε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Ευχαριστώ ο κύριος Μαλίνοφ για ένα λεπτό. Ναι, να παρέμβω κι εγώ, έστω και με καθυστέρηση. Εφόσον όλοι ε, σας επενούν, να κάνω κι εγώ έναν επενό Ψηφίσαμε το Europass σήμερα το πρωί και θυμάμαι ότι ε, μια από τις καλύτερες προτάσεις ε, αλλαγής ε, και ανανέωσης προέρχεται από τη δική σας οργάνωση. Σε γενικές γραμμές η συνάντηση με νέους ανθρώπους από αυτές τις οργανώσεις μας δίνουν μια άλλη μας δίνει μια άλλη διαφορετική προοπτική. Να σας δώσω όμως και εγώ τώρα μια άλλη προοπτική για τα προβλήματα των νέων. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας είναι ένα θέμα το οποίο δεν το συζητούμε νομίζω αρκετά. Ένα στους πέντε νέους κινδυνεύει με κοινωνικό αποκλεισμό και με φτώχεια. Ε, πάνω από ένα στους πέντε νέους ε, μεταναστεύει από την Ανατολική προς τη Δυτική Ευρώπη. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα μετά την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι είμαστε φιλοευρωπαίοι, είμαστε ενθουσιώδεις, αλλά εδώ έχουμε οκτώ ε, κράτη-μέλη της Ένωσης, ε, μεταξύ των οποίων και η Βουλγαρία, που μπορεί να μην είναι χειρότερη περίπτωση, όπου έχουμε νέους εκπαιδευμένους με δεξιότητες, ε, αυτούς που συμμετέχουν και στα φόρουμ αυτά. Αυτοί οι νέοι που η οικονομία κάθε χώρας θα ήθελε να έχει, φεύγουν. Οι πολιτικοί δεν το αναγνωρίζουν αυτό και βεβαίως δεν ζητάει κανείς τη γνώμη των νέων για αυτά. Αλλά εφόσον ε, τα συζητείτε αυτά με τις οργανώσεις στις διάφορες χώρες, είναι ένα ερώτημα που σας θέτω σε όλους σας. Αυτό το πρόβλημα δεν πρόκειται να επιληθεί εύκολα. Οποιαδήποτε όμως βοήθεια από οποιονδήποτε είναι καλοδεχούμενη. Πρωτοβουλίες, συγκεκριμένες προτάσεις, ε, συμβολικές κινήσεις, οτιδήποτε. Δεν μιλάμε γι' αυτό αρκετά. Έχω και άλλη ε, ερώτηση, αλλά θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ. Ήταν μια πολύ ε, τεταμένη ερώτηση, κύριε Γιαμάμα. Ναι, να απαντήσω πολύ ειλικρινά. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχουμε συζητήσει ως πλατφόρμα. Δηλαδή δεν έχει αποτελέσει αυτό θέμα συγκεκριμένο θέμα συζήτηση. Ταυτόχρονα συνδέεται λίγο με αυτό που είπα προηγουμένω ε, για το ότι η Ευρώπη πρέπει να συμπληρώσει τα κενά ε, με τα κράτη-μέλη. Δεν θέλω ε, βεβαίως να μπω στα χωράφια του επόμενου μιλητή, αλλά έχω συζητήσει με τον Βούλγαρο συνάδελφο που θα μιλήσει για τις επιπτώσεις τη στρατηγική για του νέου στη Βουλγαρία και νομίζω ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα ακριβώς του πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να καλύψει τα κενά και πώς μπορεί να, να βοηθήσει να δημιουργηθούν οι συνθήκες, η πρόσβαση σε δικαιώματα, οι κατάλληλες προϋποθέσεις σε εθνικό, σε τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί και αυτό το θέμα μεταξύ άλλων. Ως πλατφόρμα όμως δεν μπορώ να πω ότι το έχουμε συζητήσει ε, έως τώρα τουλάχιστον. Ευχαριστώ. Ε, υπάρχουν δύο ακόμα παρεμβάσεις ε, και θα ολοκληρώσουμε στη συνέχεια το γύρο των ερωτήσεων. Η κυρία Πόσκο. Του Κυρία Πόσκο. Τι... Ευχαριστώ. Έχουμε συναντηθεί Έχουμε συναντηθεί πολλές φορές με προσώπους ε, του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νέων ε, από το 2014 στο 2015 είχαμε την ε, εξέταση, την έκθεση μάλλον αναθεώρησης και κατά την προπαρασκευή της έκθεσής μας Ε, μπορέσαμε να συλλέξουμε εμπειρίες από τους νέους. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι χρειαζόμαστε μια στρατηγική για να αποφασίζουμε πώς μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε όλους αυτούς τους νέους που δεν συμμετέχουν σε καμία οργάνωση και πώς να τους βοηθήσουμε. Ποια όμως είναι η δική σας εμπειρία. Ε, τα κράτη-μέλη τι καλό έχουν κάνει στον τομέα αυτό που να μπορούμε και να εμπνευστούμε και εμείς. Ναι, ακούστε, ναι, μιλήστε ανοιχτά. Και ελεύθερα, λέει η Πρόεδρος. Και για τα κράτη-μέλη, δηλαδή, μπορείτε να τα πείτε ευθέως. Όχι, εγώ θα είμαι ε, ειλικρινής ε, να σας πω ότι δεν μπορώ να απαντήσω το ερώτημα αυτό, αυτή τη στιγμή. Έχουμε ενδεχομένω κάποια στοιχεία από τα μέλη μας ε, τα κράτη-μέλη αλλά δεν μπορώ να σας πω κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή για να απαντήσω. Η Σίλβια, για ένα λεπτό. Λέει πρίμα. Εσείς ε, προηγουμένως είπατε κάτι που μου άρεσε πολύ. Είπατε ότι εμείς δεν θέλουμε απλώς να εισακουστούμε για τις πολιτικές μας, δηλαδή τις πολιτικές που είναι αφιερωμένες στους νέους, αλλά να εισακουστούμε και στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Δηλαδή, ε, να μην δούμε μόνο τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη για τους νέους, αλλά ε, το γεγονός ότι χάνουμε, το ε, γεγονός ότι δεν δεχόμαστε τι μπορούν να κάνουν τα νέα παιδιά, οι φοιτητές, οι σπουδαστές για το μέλλον της Ευρώπης. Είναι κάτι που αφορά την ηθαγένεια λοιπόν και τον πρωταγωνιστικό ρόλο των παιδιών των νέων ανθρώπων. Τι θα θέλατε λοιπόν εσείς να κάνετε περισσότερο για το μέλλον της Ευρώπης, αλλά όχι ρητορικά. Υπάρχει κάτι συγκεκριμένα το οποίο και εναντίον των εθνικισμών, ε, τα τείχη που υψώνονται, το κλείσιμο. Οι ε, νέοι δεν είναι ευρωσκεπτικιστές, είναι ευρωανυπόμονοι, αυτή είναι η απόψή μου. Ε, προσπαθούν να προχωρήσουν. Δεν είναι επιφυλακτική η νέα, είναι επιφυλακτική ε, για αυτά τα οποία δεν κάνει η Ευρώπη ή ακόμα δεν είναι ακόμα η Ευρώπη. Τι θα μπορούσατε να κάνουμε λοιπόν και εμείς από πολιτική σκοπιά, ώστε να υπάρχει πλήρης ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Ε, νομίζω ότι θα χρειαστούμε ένα ακόμα απόγευμα για να καλύψουμε όλα αυτά τα σημεία ε, τα οποία ε, θα μπορούσαμε να καλύψουμε. Ως γνωρίζετε, η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης γίνεται εν μέρη και εκτός εδώ του κτηρίου. Έχουμε ευρωεκλογέ του χρόνου και αυτές είναι στιγμές ε, στις οποίες μπορούμε και θα πρέπει να θέσουμε το θεματολόγιο της νεολαίας στο προσκήνιο συζητήσαμε, εγκρίναμε τη θέση μας για το μέλλον της Ευρώπης το Μάιο, πέρσι και ήταν ένα πάρα πολύ φιλόδοξο έγγραφο το οποίο κάλυπτε όχι μόνο τομεί της πολιτικής νεολαίας αλλά και άλλους τομείς, κάλυπτε τα θεσμικά όργανα, πώς θέλουμε να έχουμε τη συμμετοχή και τη δέσμευση των θεσμικών οργάνων και αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθούσαμε να διαβιβάσουμε πολύ συχνά σε οποιοδήποτε ε, εκδήλωση που υπάρχει στο περιθώριο, στα πλαίσια ε, και τον συζητήσω με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, πώς μπορώ να τα πω όλα σε λίγα δευτερόλεπτα. Από τις οργανώσεις των μελών μας έχουμε αντιληφθεί ότι η Ευρώπη έχει πάρα πολλές δυνατότητες, οι οποίες αυτή τη στιγμή ε, δεν είναι προσβάσιμες με τον ίδιο τρόπο σε όλους. Υπάρχουν νέοι οι οποίοι αποφελούνται από προγράμματα ε, και οργανώσει νεολαία που ωφελούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα και σε γενικέ γραμμέ η αίσθηση είναι ότι αυτό είναι κάτι το εξαιρετικό. Αλλά είναι πάρα πολύ άνηση η δυνατότητα που προσφέρεται. Πολλά από αυτά τα προγράμματα, για παράδειγμα, για να αναφέρω και το Erasmus In, είναι τόσο μεγάλη ζήτηση που δεν μπορούν να καλύψουν ε, τις ανάγκες σε πολλούς τομείς, στους οποίους υπάρχουν πολύ μεγάλες ανάγκες. Ε, μπορεί να το χρησιμοποιήσει και κάποιο στο Twitter και να το πει και εκτό ε, πλαισίου. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη, υπό την έννοια ότι η Ευρώπη μας έχει ήδη υποσχεθεί ε, πολλά εμάς τη νέα γενιά. Δεν θέλουμε λοιπόν τίποτα τρελό, θέλουμε να γίνουν σεβαστές αυτές οι υποσχέσεις και να υπάρχει δυνατότητα πρόσβαση για όλου και όχι για κάποιου νέου μόνο, ένα τμήμα των νέων. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και για τη ειλικρινή σας λόγια. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Τσάμπαλη, ο οποίος εκπροσωπεί την Επιτροπή των Περιφερειών και ε, πρέπει να φύγει γιατί έχει αεροπλάνο. Θα ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Τσάμπα Μπόρμπολη πρώτα πριν να ακούσουμε τους εκπροσώπους από την Ισπανία και την Βουλγαρία. Παρακαλώ. Κύριε Μπόρμπολη, έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μια καλή ευκαιρία για μας από την Επιτροπή των Περιφερειών. Εγώ είμαι εισηγητής ε, για τα θέματα της νεολαίας και της εκπαίδευσης. Σήμερα θα μιλήσω για την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Νεολαίας από την προοπτική ε, των τοπικών και περιφερειακών πολιτικών. Με άλλα λόγια, ποιος είναι ο ρόλος ε, των τοπικών και περιφερειακών αρχών ε, για να εξασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες για όλους τους νέους ανθρώπους. Πώς ε, μπορούν να βοηθήσουν την κοινωνική ένταξη, την ενεργό συμμετοχή των νέων και τις κατάλληλες κοινωνικές πολιτικές. Πρώτον, ο στόχος της πολιτικής για την νεολαία θα πρέπει να φροντίζει να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ε, να προωθεί την κοινωνική ένταξη, να βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των νέων ανθρώπων ε, στην αγορά εργασίας, να βοηθά την ενεργό ε, ηθαγένεια να ενισχύει την έλλειψη διακρίσεων και να λαμβάνει υπόψη τη αυτά τα στοιχεία. Υπ' αυτή την έννοια όλες οι στρατηγικές για την νεολαία και οι πολιτικές περιλαμβάνουν κάποια κοινά μέτρα, κατά πολέμηση των φαινομένων των διακρίσεων ε, λόγω φυλής ή εθνοτικής καταγωγής ε, ε ή λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή αναπηρίας. Όσον αφορά την ένταξη των ε, πιο μειονεκτικών ομάδων νέων ανθρώπων, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην ένταξη αυτών των νέων ανθρώπων, ε, για παράδειγμα των λεγόμενων NEET, των ανθρώπων που δεν είναι σε εκπαίδευση, κατάρτιση ή ε, σε θέση απασχόληση και να προσφέρουν ίσες ευκαιρίες. Όσον αφορά τους ευάλωτου νέους ανθρώπους πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν σαφεί ανάγκες για πρωτοβουλίε για να υποστηρίξουν τους νέους ανθρώπους ε, που ε, εγκαταλείπουν το σύστημα μέρημνα. Θα πρέπει επίσης να μπορούμε να εγγυηθούμε ένα βασικό πακέτο για τους νέους, το οποίο θα μπορούσε να επικεντρώνεται στα εξής πέντε στοιχεία. Ε, πρόσβαση σε ε, ε, ίντερνετ γρήγορο ίντερνετ, εκμάθηση δεύτερης γλώσσας, συμμετοχή σε εθελοντισμό, πρόσβαση σε μορφές χρηματοδότησης για να μπορέσουν να κάνουν περαιτέρω σπουδές που θα τους προσφέρουν δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας από εκεί και πέρα θα πρέπει να βοηθούμε ε, την ενεργό συμμετοχή ε, των πολιτών. Η συμμετοχή των νέων ανθρώπων σε πολιτικές ε, δραστηριότητες, κυρίως όσον αφορά τη συμμετοχή και τα ποσοστά συμμετοχής στις εκλογές, είναι πάρα πολύ χαμηλά σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Παρά το γεγονός αυτό, πολλοί νέοι άνθρωποι ε, ενδιαφέρονται για τις δραστηριότητες ε, των οργανώσεων ε, της νεολαίας, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον εθελοντισμό. Και ίσως θα έπρεπε να μειώσουμε την ηλικία στην οποία μπορεί να ψηφίσει κάποιος και θα έχουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουν νέοι στη δημοκρατική διαδικασία και να εισακούγεται η άποψή τους. Οι νέοι άνθρωποι θα πρέπει να συμμετέχουν σε διαδικασίες διαμόρφωσης της κοινή γνώμης σε διάφορα πολιτικά επίπεδα ε, και σε όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς πολιτικής. Αυτό θα πρέπει να γίνει υπό τη μορφή του δομημένου διαλόγου. Για παράδειγμα, θα πρέπει να ε, συμμετέχουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές ε, στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των στρατηγικών για την νεολαία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες, ε, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι οι νέοι άνθρωποι από τις περιοχές της Υπέθρου και τις περιφέρειες πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες. Ε, πρέπει να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για νέους ανθρώπους που ζουν σε μικρούς, μικρές απομακρυσμένες κοινότητες, ε, στις εξόχους απομακρυσμένες περιοχές που αντιμετωπίζουν και δημογραφικές προκλήσεις ε, αυτές οι στρατηγικές ε, και τα προγράμματα δράσης θα πρέπει να προσπαθούν να ε, συγκεράσουν τις δεξιότητες με τις ανάγκες ε, του εργοδότη, την παραγωγή και τις ανάγκες της περιοχής. Πρέπει επίσης να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στον πληθυσμό των περιοχών της υπαίθρου που είναι στρατηγικό στοιχείο ε, πρέπει αυτοί οι νέοι άνθρωποι να δεσμεύονται για τις δραστηριότητες ε, της περιοχής της υπέστρου και η οικονομική και η κοινωνική ένταξη αυτών των ανθρώπων θα πρέπει να παρέχεται μέσω στοχευμένων προγραμμάτων και τη συμμετοχή τους. Ε, δεν χρειάζεται να τονίσουμε πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσουν εδώ οι τοπικές και περιφερειακές κοινότητες. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι αρμόδιες για την εξέβρεση των τοπικών λύσεων οι οποίες αφενών θα, βοηθήσουν ώστε η εν λόγω περιφέρεια να είναι πιο ανταγωνιστική και αφετέρου θα ενισχύσουν ε, τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των νέων ανθρώπων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ξεκινήσουμε και πάλι με την... Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε θεώρησα πολύ σημαντικό να δούμε την ε, προοπτική την τοπική και την εθνική, γιατί πολλές φορές λέμε ε, τι είναι αρμοδιότητα είναι, είναι η εθνική αρμοδιότητα, περιφερειακή, ευρωπαϊκή κλπ. Και θεωρώ ότι ερώτηση, το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να οργανωθούμε καλύτερα και πώς μπορούμε να κάνουμε ένα καλύτερο συντονισμό. Θα ήθελα να μου πείτε από περιφερειακή άποψη. Ε, τι είναι αυτό που χρειάζονται από την προοπτική των ευρωπαϊκών περιφερειών. Τι μορφή χρηματοδότησης χρειάζονται οι περιφέρειες, ούτως ώστε όλα αυτά να γίνουν πιο αποτελεσματικά. Γιατί όλοι θέλουν να συμμετάσχουν κλπ. Ποιος θα πρέπει να είναι λοιπόν ο λόγος της Ευρώπης σε αυτό το επίπεδο της περιφερειακής πολιτικής. κύριε ε, θεωρούμε, όπως είπα προηγουμένως, στο επίπεδο των αρμοδιοτήτων, θεωρούμε ότι οι νέοι θα πρέπει να έχουν πέντε δεξιότητες θα πρέπει να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για όλους τους νέους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Και θα ήθελα να συμφωνήσω με, τον, με την προηγούμενη ομιλήτρια. Ως εισηγητής για ζητήματα νεολαίας, είδα πολλά προγράμματα που να σχετίζονται με την ε, εγγύηση για την νεολαία που τελικά καρποφόρησαν. Δεν λαμβάνουμε υπόψη το γεγονός ότι αποφάσεις που επηρεάζουν τους νέους ανθρώπους θα πρέπει να λαμβάνονται σε τοπικό επίπεδο σε σχέση με τον αθλονισμό, την ε, ψυχαγωγία κλπ. και άλλες ε, ευκαιρίες σε τοπικό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή ε, επεξεργαζόμαστε μια έκθεση για την εκπαίδευση. Το πρόγραμμα Erasmus δεν αρκεί. Θα πρέπει να εξετάσουμε και άλλα αναπτυξιακά προγράμματα, ούτε ώστε να είμαστε σε θέση να παράσχουμε τους... να έχουν οι νέοι άνθρωποι κάποια αποθέματα γιατί μόνο σε χώρες όπου ε, έχουν ε, λειτουργήσει, δουλέψει κάποια προγράμματα, οι νέοι ε, έχουν τύχει κάποιας προσοχής. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα πρέπει επίσης να αλλάξουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων γιατί συχνά υπάρχουν 50 ή 100 σημεία στην ημερήσια διάταξη χωρίς κανένα από αυτά να αφορά τους νέους ανθρώπους. Θα πρέπει να αλλάξει αυτή η 100 σημεια στην ημερησια χωρις κανενα απο αυτα να αφορα τους νεους ανθρωπους θα πρεπει να αλλαξει αυτη η κατασταση και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις τοπικές αλλά και τις εθνικές πολιτικές οι οποίες γενικά λαμβάνουν ε, μέτρα οι πολιτικές για ανθρώπους που είναι ψηφοφόροι. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω να υπάρχουν άλλες ε, παρεμβάσεις. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά. Εάν πρέπει να αποχωρήσετε, ε, δεν θα σας παρεξηγήσουμε. Και, αλλά περιμένουμε με ανυπομονησία την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειών και ελπίζουμε ότι και εσείς θα, πάρετε κάποιο, θα πήρατε κάποιο ερέθισμα από τη σημερινή συζήτηση που θα συμπεριλάβετε στην εκθεσή σας. Ωραία. Τώρα θα έρθουμε στον κύριο Ντένι Σιτάσο, ο οποίος είναι βουλευτής αρμόδιος για τουρισμό, αθλητισμό και πολιτισμό ε, σε μια περιοχή της Ισπανίας. Έχει το λόγο για 10 λεπτά. Eh, Eh, Ευχαριστώ πολύ. Να σας πω ότι λέγομαι Ντενίση Τσάσο, είμαι υπεύθυνο πολιτισμού, νεολαίας και αθλητισμού στην περιοχή του Σαν Σεμπαστιάν, σε μια επαρχία της χώρας των Βάσκων στην Ισπανία και να ευχαριστήσω και την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μας έδωσε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε σε αυτή τη δημόσια ακρόαση για τη στρατηγική για την νεολαία. Ερχόμαστε εδώ να σας παρουσιάσουμε την εμπειρία μας ε, για ε, την ψηφιακή κουλτούρα. Η ψηφιακή επανάσταση, το διαδίκτυο, ε, αλλάζει πολλές πτυχές της ζωής μας. Καταρχάς την επικοινωνία, την ενημέρωση, τα οικονομικά, τη σχέση μεταξύ των ανθρώπων, την ψυχαγωγία, τη διασκέδαση, τις μεταφορές, την πολιτική συμμετοχή και πολλούς άλλους τομείς, στους οποίους οι νέοι και οι νέες έχουν πολλά να πούνε και θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα τμήμα της κοινωνίας ε, που αφορά τους νέους, ε, που είναι ιδιαίτερα ευάλωτο για, ε, ενώπιον των κινδύνων του ψηφιακού κόσμου και της εποχής του διαδικτύου. Να πω ότι είναι ένας τομέας ο οποίος είναι γεμάτος ευκαιρίες και μα επέτρεψε να προοδεύσουμε ω κοινωνία, αλλά σε κανέναν δεν διαφεύγει το γεγονό ότι είναι και γεμάτο κινδύνους. Και γιατί για τους νέους. Πιστεύουμε ότι ο κόσμο των νέων και των εφήβων ε, περιλαμβάνει πάρα πολλά κίνητρα ε, λόγω των εξωτερικών ε, εμπειριών και ερεθισμάτων και λόγω του διαδικτύου και δεν έχουν και την εμπειρία που έχουν ίσως και κάποιοι ενήλικες που ορισμένε φορές περνάνε ίδια μια διαδικασία εκμάθησης και προσαρμογή σε όλα αυτά. Το πρόγραμμα της ε, ψηφιακής κουλτούρας, το κουλτούρα digital όπως λέγεται, τέθηκε σε εφαρμογή με σκοπό να εκπαιδεύσουμε ε, για κατάλληλη χρήση των νέων τεχνολογιών, αλλά και προσπαθούμε και να ε, σπάσουμε αυτό το χάσμα γενεών και το εδαφικό χάσμα που δημιουργείται όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες. Και πιστεύουμε ότι αυτή η στρατηγική για την ψηφιακή εκπαίδευση, τον ψηφιακό πολιτισμό, περιλαμβάνεται στα όσα προβλέπουμε ...επί το σχέδιο και η στρατηγική για την νεολαία που συζητάτε τώρα και που προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες ε, για ε, τα ψηφιακά δίκτυα. Να μπω στο προκείμενο, να σας πω ότι αυτό το ε, πρόγραμμα, το Cultura Digital, περιλαμβάνει τρεις πτυχές η πρώτη έχει σχέση με την μάχη κατά του cyberbullying. Όλοι γνωρίζετε ότι το bullying, όπως και άλλες κοινωνικές παθήσεις, έχει και τη δική του διάσταση στο διαδίκτυο και κυρίως έχει ένα πολλαπλασιαστικό παράγοντα ε, στη ε, ζημιά που μπορεί να προκαλέσει στο νέο ή στο θέμα. Ε, και υπάρχει ένα άλλο σκέλος, προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε καλύτερα στους νέους ανθρώπους αυτή τη γλώσσα που είναι όλο και πιο σημαντική και θα είναι και στο μέλλον πολύ πιο σημαντική για να μπορούν να κρίνουν και να είναι και ικανοί να ασχολούνται με τον κόσμο του διαδικτύου, γλώσσες προγραμματισμού δηλαδή. Και υπάρχει και το Instant Batean που είναι ένα άλλο πρόγραμμα στο οποίο ε, έχουμε ε, μια δυνατότητα ανταλλαγών ε, μεταξύ νέων Βάσκων με άλλες περιοχές της Ευρώπης, εργαστήρια καλοκαιρινά, θερινά εργαστήρια για τα πλεονεκτήματα και τις προκλήσεις που έχει ο κόσμος του διαδικτύου όσον αφορά την διασκέδαση και την ψυχαγωγία και κατάρτιση στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus Sin για τους ε, τεχνικούς, τους επαγγελματίες που πρέπει να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις προκλήσεις και να μπορέσουν να εκπαιδεύσουν τους νέους μας ε, ε, σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία ε, σχετίζονται με το διαδίκτυο. Τώρα, για το πρώτο λοιπόν από τις ενότητες, το cyberbullying, τον εκφοβισμό δηλαδή στο διαδίκτυο, αυτό το οποίο καταφέραμε να κάνουμε μαζί με, την, με το Πανεπιστήμιο της χώρας των Βάσκων, καταφέραμε να έχουμε ε, υλικό το οποίο δίνει τη δυνατότητα και στους εκπαιδευτικούς αλλά και ε, στους γονείς ε, να μπορούν να διαπιστώσουν εγκαίρως περιστατικά cyberbullying. Υπάρχει το πρόγραμμα FisherNet το οποίο εκπαιδεύει μέσω ομάδων έρευνας άτομα τα οποία μπορούν να κάνουν προτάσεις ε, δράσεις ε, στους νέους, ε, στους εφήβους και το πώς μπορούν να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες και επίσης υπάρχουν και διάφοροι διάλογοι και εργαστήρια ε, στην περιοχή μας ε, με τον ίδιο σκοπό, να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε και να δώσουμε γνώσεις και πληροφορίες για τους κινδύνους ε, και την πραγματικότητα αυτή του cyberbullying και η οποία πολλές φορές είναι και καλυμμένη μέχρι να υπάρξει κάποιο περιστατικό, μέχρι να φτάσουμε στην θλιβερή πραγματικότητα. Περνάμε στο δεύτερο σκέλος αυτού του προγράμματος του ψηφιακής εκπαίδευσης, λέγεται Code και όπως σας είπα προηγουμένως, ε, λαμβάνουμε υπόψη μας ότι οι γλώσσες προγραμματισμού, ε, ο κώδικας είναι μια παγκόσμια γλώσσα ε, και θα κυριαρχήσει στο η χρήση της τεχνολογίας και εδώ υπάρχουν κάποια κενά εδαφικού χαρακτήρα. Προηγουμένως αναφερθήκαμε στην αναφορά του κόσμου της υπαίθρου και του άστεως. Υπάρχει χάσμα γενεών και υπάρχουν και χάσματα λόγω του οικονομικού επίπεδου των οικογενειών. Και επομένω θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα κενά, ώστε κάθε νέος, ανεξάρτητα από τις προσωπικές του συνθήκες, να έχει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε αυτές τις γνώσεις, οι οποίες θα είναι βασικέ γνώσει, όπω το παρελθόν ήταν να γνωρίζει κάποιος να διαβάζει, να γράφει κλπ. σε αυτή τη ε, πτυχή έχουμε κάνει διάφορες δραστηριότητες, ε, υπήρχαν ε, τεχνολογικές, τεχνολογικά εργαστήρια σε επιχειρήσεις που είναι τεχνολογικές επιχειρήσεις, γίνονται στις σχολικές διακοπές και τη Μεγάλη Εβδομάδα και τα Χριστούγεννα. Ε, ίσως η πιο αξιοσημείωτη δραστηριότητα που είχε και το μεγαλύτερο αντίκτυπο στην περιοχή ήταν ένα λεωφορείο ε, το οποίο ε, ήρθε και με χορηγία μιας ε, τοπικής επιχείρησης που κατασκευάζει λεωφορεία, το οποίο κυκλοφόρησε σε διάφορες περιοχές της επαρχίας, μετέφερε πάνω από χίλιους νέους σε διάφορες περιοχές και έγιναν εργαστήρια προγραμματισμού ο οποίος προγραμματισμός είναι και το αντικείμενο αυτής της ενότητας του κόντε του. Είχαμε θερινές διακοπές ε, ψηφιακές σε διάφορες περιοχές, εκμεταλλευτήκαμε και ε, τους διάφορους ξενώνες ε, που έχει η περιοχή. Υπήρχε και ένα πάρκο Χριστουγέννων σε ένα δήμο, στον οποίο συμμετείχανε ε, περίπου 300 νέοι. Και τέλος υπάρχει η δραστηριότητα Instant EAN που αναφέρεται σε φίβους ε, για να προλάβουν τους κινδύνους των νέων τεχνολογιών. Προσπαθεί να προστατεύσει από τον ε, ψηφιακό κόσμο και να γίνεται διάκριση μεταξύ πραγματικού και ψηφιακού κόσμου. Προσπαθούμε να δούμε τις διαφορές μεταξύ ψηφιακού και πραγματικού κόσμου με πράγματα τα οποία μπορούν να διαπιστώσουν οι ενήλικες. Είναι αλήθεια ότι το διαδίκτυο είναι ένας κόσμος ε, χωρίς ε, τύχη, χωρίς πόρτες, ε, μπορεί να υπάρχει οποιοδήποτε περιεχόμενο ε, που ορισμένες φορές μπορεί να είναι και δύσκολο ε, να διακρίνει κανείς μεταξύ του πραγματικού και του φανταστικού και ίσως ε, θα πρέπει να υπάρχει και εκπαίδευση, να μάθουν τα παιδιά τις κατάλληλες αξίες και να αναπτύξουν και κριτική ικανότητα, να θέσουν ερωτηματικά και να μπορέσουν να αναρωτηθούν από πού λαμβάνουν συγκεκριμένες πληροφορίες, από ποιες πηγές και να έχουν και την κριτική ικανότητα να αντιληφθούν τις πληροφορίες που βρίσκουν στο διαδίκτυο. Να υπάρχει λοιπόν δυνατότητα κριτικής ικανότητας και να προσφέρουμε και δυνατότητες ε, κατάλληλης συμπεριφεράς ε, και ε, αγωγής του πολίτη μέσω του διαδικτύου. Μέσω αυτού του προγράμματος του Ισταντεάν ε, είχαμε πάλι εργαστήρια, διαγωνισμούς φωτογραφίας και βίντεο στο Instagram και ε, διάλογο με YouTubers, με ανθρώπους οι οποίοι κάνουν βίντεο στο YouTube. Και επίσης είχαμε και συμμετοχή με το Erasmus Sim. αυτό το οποίο κάναμε ε, ήταν να έχουμε συγκεκριμένε συναντήσει που έγιναν τον Οκτώβριο του 2017 μεταξύ νέων και επαγγελματιών, ε, εμπειρογνωμόνων της περιοχής, ε, με πόλεις επίσης όπως το Μπισμπάντεν, στη Σλοβενία, πόλεις της Τουρκίας και του Ισραήλ. Για να έχουμε ευκαιρίες και κινδύνους για τον ψηφιακό κόσμο, για να μπορέσουμε να εργαστούμε με εφήβους και νέου. Και τέλος, σε αυτή την ενότητα του Erasmus Sin, Έχουμε το Inno Youth, στο οποίο συμμετείχαν ε, ε, οι δήμοι της περιοχής μας. Ε, είχαμε συμμετοχή του Δήμου της Βεργάρα και του Βισβάντεν και έγινε το Σεπτέμβριο το Σεπτέμβριο στην χώρα των Βάσκων και τον Οκτώβριο στη Γερμανία και είχε σχέση και με την καθημερινότητα των νέων. Αυτά λοιπόν είναι η πιο συγκεκριμένη εμπειρία και πρόταση που είχαμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρακτική ε, ματιά που μας δώσατε στην εργασία αυτή που γίνεται για τους νέους και πήραμε μία ιδέα για το πώς μπορούμε να προωθήσουμε την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων για τους νέους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έχει υποβάλει ένα πρόγραμμα δράση, εκπονεί ένα πρόγραμμα δράση, γι' αυτό είναι πολύ χρήσιμο ε, να δούμε πώς μπορεί να είναι μια τέτοια βέλτιστη πρακτική, ούτως ώστε να αντλήσουμε κάποια καλά στοιχεία από αυτό το παράδειγμα. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε πολύ. Ε, Ευχαριστώ πολύ, όπως είπε και η Πρόεδρος. Είναι αλήθεια ότι για τα ζητήματα αυτά έχουμε μιλήσει πολύ σε αυτή την Επιτροπή. Αυτό που θα με ενδιέφερε εμένα είναι αυτές οι τοπικές εμπειρίες, ε, διότι όντως το ίντερνετ ε, έχει κατά κάποιο τρόπο εισβάλλει στις ζωές μας πότομα Έχουμε όμως και ε, άλλα, άλλους τρόπους εμείς ε, οι παλαιότεροι για να ε, αμυνθούμε απέναντι σε τέτοιου είδου ε, ειδήσει, ενώ οι πιο νέοι λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες χωρίς κανένα φιλτράρισμα. Θέλει λοιπόν προσοχή. Ταυτόχρονα το διαδίκτυο έχει και ένα άλλο ε, κρυφό ε, αποτέλεσμα ότι δημιουργεί νέους αναλφάβητους. Σε θεσμικό λοιπόν επίπεδο τι γίνεται ε, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό τομέα για, το πώς θα, για, να μπορέσουμε να μετριάσουμε αυτές τα δύο ε, αρνητικά στοιχεία. Δηλαδή το μη φιλτράρισμα του περιεχομένου και ε, οι δεξιότητες οι οποίες χάνονται στον ψηφιακό κόσμο. Ναι, ευχαριστώ Έιντερ. Εγώ θεωρώ, πόσο ξέρω τουλάχιστον, το εκπαιδευτικό σύστημα δίνει δυνατότητες σε τεχνικό επίπεδο στους νέους και στις νέες. Όμως αυτό που μας λείπει, το μόνιμο πρόβλημα, η μόνιμη πρόκληση της κάθε του κάθε εκπαιδευτικού συστήματος είναι η δημιουργία κριτικής σκέψης. Να μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει κάποια πράγματα σε μια εποχή ε, μετααλήθειας ε, εμείς έχουμε συνηθίσει περισσότερο ενδεχομένως ή ε, ενδεχομένως να έχουμε κληρονομήσει ε, κάποια πράγματα από ένα σύστημα το οποίο καταλάβαμε καλύτερα, καταλάβαμε καλύτερα τις διαφορές. Τη σήμερα ημέρα όμως, ε, πατώντας ένα κουμπί, μπαίνει κάποιος σε οποιαδήποτε σελίδα στο διαδίκτυο, λέγοντας απλώς ότι είναι 18 χρονών, χωρίς να το ελέγχει κανείς, και εκεί μπορεί να προωθούνται ε, αρνητικές αξίες, ε, αξίες ε, οι οποίες μπορεί να πηγαίνουν σε βάρος, να πλήττουν την εικόνα της γυναίκας, τους ανθρώπους με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, με διαφορετικό κοινωνικονομικό υπόβαθρο. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι είναι αναγκαίο να εκπαιδεύσουμε τους νέους ώστε να αποκτήσουν την κριτική αυτή σκέψη, να επαληθεύουν, να τσεκάρουν, αν θέλετε, τις πηγές των ειδήσεων. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Σαρόβα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσίασή σας γιατί είστε εκπρόσωπος της περιφερειακής κυβέρνησης, δηλαδή ενός κοινοβουλίου. Και εμένα θα με ενδιέφερε να μας πείτε κατά πόσο το project αυτό με, την, με μια ε, έγινε σε συνεργασία με, τοπική, με την τοπική διοίκηση ήταν μια πρωτοβουλία των ερετών. Ε, εν πάση περιπτώσει είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα ε, και πιστεύω ότι υπάρχουν πράγματι ελλείμματα ε, κριτικής σκέψης και αυτό υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρώπη και είναι και ένα θέμα παιδαγωγών. Υπάρχουν πολύ λιγοστοί ε, δάσκαλοι, καθηγητές οι οποίοι θα ήταν διατεθειμένοι να εργαστούν στην κατεύθυνση αυτή. Ε, άρα θα πρέπει αυτό να αντικατασταθεί με εξωσχολικές, ε, από εξωσχολικές δραστηριότητες και συνιστά βεβαίω μια για, ε, πρόκληση για οργανώσεις νέων. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ για το ερώτημα. Πρέπει να πω ότι ήταν πολιτική η όθηση που δόθηκε την πρωτοβουλία αυτή και έχουμε εδώ τη διευθύντρια, την υπεύθυνη ε, για αυτό το θέμα είναι και μητέρα τριών παιδιών και ζει αυτή την πραγματικότητα καθημερινά και ίσως γι' αυτό να έδωσε και τόση όθηση. Διαπιστώνουμε επίσης γύρω μας ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, το είπατε κι εσείς πολύ σωστά, υπάρχει ένα πρόβλημα του κατά πόσο οι επαγγελματίες του κλάδου, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί, έχουν τα κατάλληλα εργαλεία, έχουν τις κατάλληλες γνώσεις για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτή τη νέα πραγματικότητα. Είχαμε πετύχει οι καθηγητές αυτοί σιγά σιγά να ε, συνειδητοποιήσουν τη νέα πραγματικότητα, ε, παραδείγματο χάρη ό,τι αφορά το bullying. όμως ο πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα ε, ε, μέσω των κινητών τηλεφώνων, ε, όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία αυξάνουν την πίεση ε, προς το θύμα, ε, πραγματικά ορισμένες φορές έχει καταλυτικά αποτελέσματα, ολέθρια για κάποιον που υφίσταται αυτή την πίεση. Πρέπει λοιπόν να μπορούν και οι καθηγητέ ε, και το εκπαιδευτικό προσωπικό να μπορούν να κινηθούν στο διαδίκτυο, να ξέρουν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία αυτά. Και εκεί είναι που πρέπει να γίνει μια προσπάθεια. Ευχαριστώ κύριο ε, Ζάμιτ Ντίτριχ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για την παρουσίαση. Δώσατε έμφαση στο κυβερνομπούλινγκ και στην εκπαίδευση των νέων ανθρώπων σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό, αλλά ένα από τα βασικά προβλήματα νομίζω ε, είναι ακριβώς η δυνατότητα ανάπτυξης κριτικής σκέψης. Ε, να μπορεί δηλαδή κάποιος να διαχωρίσει το τι είναι αλήθεια, τι είναι πραγματικότητα και τι είναι ψέμα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε υπερφόρτωση πληροφοριών ε, στο Google ψάχνουμε πληροφορίες, αλλά μετά πρέπει να γίνει μια επιλογή, ένα ξεσκαρτάρισμα. Ποια ε, ε, πηγή είναι αξιόπιστη και ποια όχι, όπως το Wikipedia παραδείγματος χάρη. Ε, είναι σημαντική αυτή η ανάπτυξη των, των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης. Πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες είναι πιο ευάλωτες ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Ναι, το ερώτημα είναι εξαιρετικά εύστοχο. Πριν από τρεις μέρες στο Μπιλμπάο έγινε μια επίθεση βίαιη προς ε, δύο ηλικιωμένους ε, ε, στο σπίτι τους και συνελήφθησαν τρεις νέοι ανήλικοι οι οποίοι όχι μόνο έκλειψαν τους ηλικιωμένους αυτούς αλλά τους έδιραν κιόλας άσχημα. Όταν λοιπόν αυτοί οι νέοι βλέπουν το κουριστό πορτοκάλι του Στάνλε Κιούμπρικ, πούμε, πρέπει να μπορούν να διαχωρίσουν την πραγματικότητα από την ε, ε φαντασία, ότι εδώ δεν είναι ε, μία ε, πρακτική που πρέπει κάποιος να μιμηθεί ε, στις ταινίες αυτές. αυτό που πρέπει να γίνει στο διαδίκτυο είναι οι νέοι να αντιληφθούν ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας αναπαράστασης ή ε, κάποιας ε, ταινίας και μιας πραγματικότητας και μιας πραγματικής συμπεριφοράς που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι μεταξύ τους σεβόμενοι μεν τους δε. Ε, βεβαίως ε, συμφωνώ ότι πρέπει να επιμείνουμε ε, έτσι ώστε να μπορούν οι νέοι να εντοπίσουν τις διαφορές αλλά υπάρχουν και όρια. Δηλαδή οι νέοι, όσο πιο νέοι είναι, και δεν έχουν αναπτύξει επαρκή, επαρκείς δεξιότητες για να κάνουν τη διαφορά, να υπάρχει ένα όριο, μια, ε, ένα όριο που να μην τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση σε κάποια περιεχόμενα. Αν κάποιος δώσει ένα παιδί 4 ετών ένα τάμπλετ και αρχίζει να βλέπει ένα κανάλι, να βλέπει ταινίες, βίντεο, μπορεί αυτό το παιδάκι να πατάει τα κουμπιά και να φτάσει κάπου αλλού σε ένα μέρος που δεν ελέγχουμε. Πιστεύω ότι υπάρχει, αυτή, υπάρχει τεχνολογία αυτή τη στιγμή που μας επιτρέπει να πλαισιώσουμε κάπως ε, ε, το περιεχόμενο στο οποίο έχουν πρόσβαση οι ανήλικοι, έτσι ώστε τέτοιου είδους ε, περιεχόμενα επικίνδυνα να φτάσουν σε εμά όταν είμαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος ομιλητής στο γύρο αυτό. Ωραία, λοιπόν. Άκουσα προσεκτικά και έχετε εστιάσει σε ένα διαφορετικό σημείο. Αλλά παρόλα αυτά θα ρωτήσω το ίδιο ερώτημα. Δεν βλέπω το λόγο να το αλλάξω. Απλώς θα το αναδιατυπώσω. Στην δική σας ε, περιοχή έχετε προβλήματα με υπερβολικά ε, πολλούς ε, νέους που να φεύγουν για μεγαλύτερες πόλεις γιατί τα όσα είπατε είναι πράγματι πολύ καλές πρακτικές, αλλά αν έχετε τέτοιου προβλήματα, ελπίζω όχι, αλλά αν τα έχετε, σκεφτήκατε ποτέ ε, συγκεκριμένες πολιτικές πρωτοβουλίε για να κρατήσετε τους νέους ανθρώπους στις περιοχές, στα χωριά τους, ειδικέ πρακτικές, όπως για παράδειγμα ε, νέους ε, κανόνες για την ενοικίαση ε, κινήτων, και λοιπά Γιατί η προοπτική των νέων αφορά τα δικαιώματά τους, τις ελευθερίες τους και τις ευκαιρίες τους. Αλλά όλοι γνωρίζουν τι συμβαίνει σε μια περιοχή η οποία εγκαταλείπεται από τους νέους. Ε, τίποτα ε, το καλό δεν μπορεί να συμβεί σε αυτές τις περιοχές και ίσως ε, δεν είναι... Ε, ίσως το έχετε συζητήσει αυτό. Βεβαίως μπορούμε να μετακυλήσουμε το φορτίο στις εθνικές κυβερνήσεις και να πούμε ότι θα έπρεπε να κάνουν ό,τι μπορούν. Αλλά διορτώμε κατά πόσο έχει αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Ίσως το παρελθόν, ενώ όχι τώρα. Ίσως το έχετε επιλύσει, δεν ξέρω. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, ε, ερώτηση, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να κάνω ένα σχετικό σχόλιο. Η, στην Ισπανία, η Ισπανία υπέφερε πάρα πολύ από την τελευταία χρηματοπιστωτική κρίση και γι' αυτό οδήγησε σε μια θλιβερή έξοδο των νέων και διαρροή ε, ταλέντων και ε, ε ανθρώπων προς άλλες χώρες. Στη χώρα των Βάσκων αυτή η φυγή των ταλέντων ε, νέων που δεν ε, βρήκαν αρκετές ευκαιρίες ε, στη δική τους περιφέρεια, επειδή ο αντίκτυπος της κρίσης ήταν ίσως τις πιο βιομηχανικές περιοχές της Ισπανίας ήταν μεγάλος, αλλά ίσως όχι ως άλλες περιοχές. Και υπάρχει το φαινόμενο πιο ελκυστικών ε, προσφορών ε, συμβολέων προς τους νέους αυτούς αυτή τη στιγμή τους ώστε να προσελκυστούν οι νέοι να επιστρέψουν ε, στην πατρίδα τους. Υπάρχουν λοιπόν ειδικά συμβόλαια και στη δική μας περιοχή δεν υπήρξε με τόσο έντονη ε, μορφή, σε τόσο έντονη μορφή η έξοδος αυτή την οποία βίωσαν ωστόσο άλλες ε, περιοχές της Ισπανίας. Ωραία λοιπόν. Ένα λεπτό. Ε, δεν ξέρω αν κατάλαβες τη διαδικασία. Ένα λεπτό η ερώτηση και μετά η απάντηση. Όπως και η ερώτηση του κυρίου Μαρίνοφ, να κάνω κάτι αντίστοιχο. Αναφερθήκαμε σε στόχους, ε, περιοχές των συνόρων, ιδιαίτερα την περιοχή του Ερούν, γιατί στο σχέδιο εδώ δεν αναφέρεστε, για παράδειγμα, ε, τόσο πολύ στη Γαλλία, αναφέρεστε στην ε, χώρα των Βάσκων. Υπήρξε συνεργασία σε περιοχέ, με περιοχές του Βορρά. Ξέρουμε ότι ο πολιτισμός, ο Βάσκικος είναι πάρα πολύ καλός. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία εκεί και φαντάζομαι ότι οποιοδήποτε θα μπορούσε να συμφωνήσει. Αλλά τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχουν πάρα πολλέ επαφέ, ε, πολύ μεγάλη κινητικότητα στα σύνορα, ε, πολλά συμφέροντα και από πλευρά στην χώρα των ε, Βάσκων, αλλά και πέραν των σύνορων με τη Γαλλία, πώ γίνεται η σχεση γαλλια Γαλλίας-Ισπανίας και χώρα των Βάσκων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σα λόγια και για την ερώτηση. Πρέπει να αναγνωρίσω ότι συγκεκριμένα στο πρόγραμμα αυτό δεν υπήρξε διασυνοριακή εμπειρία. Το τμήμα βέβαια της περιοχής μας έχει πολλές εμπειρίες σε θέματα τουρισμού, σε θέματα πολιτισμού και αθλητισμού. Ασχολούμαστε πολύ. Εδώ σε αυτό το θέμα δεν υπήρχε διασυνοριακή συνεργασία με την ε, περιοχή της Νότιας Γαλλίας που βρίσκεται στα σύνορά μας, αλλά υπήρχαν ε, ανταλλαγές ε, με αδελφοποιημένες πόλεις, όπως για παράδειγμα την περίπτωση του Βισμπάντεν, όπως σας παρουσίασα προηγουμένως, και άλλες πόλεις από άλλες χώρες ευρωπαϊκές ε, διότι το πρόβλημα έχει και ευρωπαϊκή διάσταση προφανώς ε, και όπως και να έχει θεωρούμε ότι η Ευρώπη είναι ο πλέον κατάλληλος χώρος για να εκπαιδεύσουμε και να ε, καταρτήσουμε τους νέους μας, να τους επιμορφώσουμε για αυτούς τους κινδύνους που είναι κοινοί για όλους. Ευχαριστώ. Αυτό ήταν ένα ρεύσμα για τη συνέχιση αυτού του προγράμματος το οποίο θα μπορούσε να προσλάβει μια διασυνοριακή διάσταση με τις ε, γαλλικές ε, ε, κοινότητες από την άλλη πλευρά των συνόρων γιατί ορισμένες φορές τα καλά πράγματα βρίσκονται πολύ κοντά δεν χρειάζεται να προσέξουμε σε απομακρυσμένες χώρες Καταρχήν σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρουσιάσετε εδώ αυτό το πρόγραμμα και τώρα θα έρθουμε στην τελευταία μας προσκεκλημένη, την κυρία Λένκοβα, Λίλια Λένκοβα, η οποία είναι τεταλμένη για το διαρθρωμένο διάλογο στο Εθνικό Φόρουμ Νεολαίας στην Βουλγαρία. Και εσείς θερμά καλώς ήρθατε και έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας για την παρουσίασή σας. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την ε, δυνατότητα να σας ε, μιλήσω. Εδώ και δέκα χρόνια εργάζομαι σε μια μη κυβερνητική οργάνωση για την νεολαία και κάνω και μια διατριβή για το θέμα της πολιτικής για την νεολαία στη Βουλγαρία. Η παρουσίασή μου θα είναι πολύ συγκεκριμένη και συστηματική. Θα διαφέρω την παρουσίασή μου σε τρία τμήματα. Καταρχήν με σύντομα παραδείγματα για το πώς οι ευρωπαϊκές πολιτικές και η σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Βουλγαρίας είχε θετικά αποτελέσματα. Πρώτον, η δημιουργία μιας μεγάλης πλατφόρμας για τους νέους στη Βουλγαρία, το Εθνικό Φόρουμ για τη Νεολαία και μπορώ να σας ότι τρεις παράγοντες επηρέασαν αυτή την εξέλιξη. Πρώτον, η επιθυμία των ε, οργανώσεων νεολαίας που είναι μέλη σε αυτή την ε, πλατφόρμα να συμμετάσχουν. Δεύτερον, η πολύ θετική εμπειρία ε, που είχαν και εξαιρετικά καταρτισμένοι νέοι leader εκεί ε, επικεφαλής. Και θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό ε, σχετίζεται άμεσα με το πρόγραμμα νεολαία δράση στη Βουλγαρία. Και ε, τρίτον ήταν η απλοποίηση του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την Νεολαία. Ευθύς εξ αρχής το φόρουμ αυτό είχε το όραμα να αποτελέσει τμήμα του Μεγάλου Ευρωπαϊκού Φόρουμ και ε, η δημιουργία ενός μιας ε, δεξαμενής ε, εκπαιδευτών. Η πρώτη γενιά πολιτικών είδε ξεκάθαρα ότι θα πρέπει να, να, λειτουργήσει, να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά όσον αφορά τη διάδοση των ευρωπαϊκών αξιών. Άρα λοιπόν εκπονήθηκε ένας ε, μηχανισμός για τον ε, πολλαπλασιασμό αυτών των ευρωπαϊκών αξιών και αυτή τη στιγμή το Εθνικό Φόρουμ για την Νεότητα σε τοπικό επίπεδο έχει εφαρμόσει σημαντικά εκπαιδευτικά μέτρα σε συνεργασία με 10 τοπικές κοινότητες ε, έγινε αυτό τα τελευταία δύο χρόνια, τα θέματα δημοκρατίας, συμμετοχή των νέων. αρμοδιότητες των νέων ανθρώπων και άλλα θέματα. Ένα από τα σημαντικά αποτελέσματα είναι η συμμετοχή του Εθνικού Φόρουμ για την Νεολαία στην Διεθνή Ομάδα Εργασίας για το Διαθρωμένο Διάλογο. Το 2014 η Εθνική Ομάδα οργασίας του Εθνικού Φόρουμ ε, εξέλεξε μάλλον, συγγνώμη, το Εθνικό Φόρουμ, η Διεθνής Ομάδα Εργασίας εξέλεξε το Εθνικό Φόρουμ ε, ως επικεφαλής και ε, διαπιστώθηκαν ε, τρεις ε, βέλτιστες πρακτικές δόθηκε πράσινο φως για τη συμμετοχή των νέων ανθρώπων σε τοπικό επίπεδο ε, και εκπονήθηκαν ε, εκπαιδευτικές διαδικασίες στο πλαίσιο του διαφερμένου διαλόγου. Τρίτον, έχουμε και μία διαδικασία για τους νέους ε, εντεταλμένους ε, που εκπροσωπούν τη Βουλγαρία στο Διεθνές ε, Φόρουμ για την Νεολαία. Αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό σε εταιρική σχέση και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής η δημιουργία μιας άμεσης εταιρική σχέσης μεταξύ του, της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Νεολαία και, την, ε, και της δικής μας ομάδας εργασίας για την Νεολαία. Και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να απαντήσω μια, οποία μια ερώτηση η οποία τέθη προηγουμένως, δηλαδή τι ε, πώς συνέφερε ο διαδρομένος διάλογος ε, στη Βουλγαρία και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι μέσω του διαδρομένου διαλόγου οι νέοι άνθρωποι από αντικείμενο της ε, πολιτικής έγιναν υποκείμενα πολιτικά γιατί πράγματι συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και λίγο πριν οι πολιτικοί εκπώνησαν ε, απλώς εκπονούσαν συγκεκριμένα εργαλεία ενώ οι νέοι ήταν απλώς οι χρήστες αυτών των πολιτικών αλλά η κατάσταση αυτή άλλαξε ριζικά Και κάτι άλλο. Πρόκειται για μια κοινοτική πολιτική, την πολιτική της πόλης της Βάρνας και τις ε, οργανώσεις νέων εκεί. Η Βάρνα έγινε η Ευρωπαϊκή ε, Πρωτεύουσα των Νέων το 2014 και είναι η μόνη πόλη η οποία έχει συγκεκριμένο προπολογισμό για τις ε, πρωτοβουλίες των νέων. Δηλαδή όχι μόνο κάτω από την ομπρέλα του αθλητισμού, του πολιτισμού ή άλλων τομέων, Και κάτι που ίσως ακούτε για πρώτη φορά ε, το σύστημα μεταφοράς ε, πιστώσεων στον εκπαιδευτικό τομέα. Εδώ έχουμε διάφορες ε, εταιρικέ σχέσεις και υπάρχει και ένα αντίστοιχο εργαλείο που είναι σύσταση της Ευρωπαϊκής Στατικής, EQUIT, ως ε, εργαλείο για την ε, πιστοποίηση αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο της άτυπης ε, εκμάθησης. Βρισκόμαστε τώρα σε μια δεύτερη φάση αυτού του προγράμματος και στοχεύουμε στο να δώσουμε στους νέους ανθρώπους τη δυνατότητα να βρουν εκεί ε, τη θέση τους και να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους ούτως ώστε η αναγνώριση των ικανοτήτων τους και ο επαγγελματικός προσανατολισμός ε, να ε, βελτιστοποιηθούν. Και τώρα θα περάσω άμεσα στο ερώτημα για τη λεγόμενη ψυχική υγεία των νέων. Και εδώ έχουμε λάβει πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Και θα ήθελα, σε σχέση με τόσο είπαν οι συνάδελφοι, να πω ότι ένα σημαντικό θέμα στη Βουλγαρία είναι η ριζοσπαστικοποίηση των νέων ανθρώπων. Και εδώ ασχολούμεθα σοβαρά με τις επαφές μεταξύ των ε, νέων, των ομιλίκων και την ένταξη στην κοινωνία ως ε, τρόπο αποφυγής του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι συγκεκριμένες συστάσεις, οι οποίες θα ήθελα να απευθύνω στην, προσεχή, στην επόμενη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τους Νέους, θα διατυπωθούν και γραπτά και αφορούν σε ορισμένα θέματα και θα επανέλθω στο πρώτο παράδειγμα λέγοντας ότι χρειαζόμαστε ένα ξεκάθαρο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για, τις, ε, για τους πολιτικούς, για την νεολαία και τη συμμετοχή των νέων ανθρώπων γιατί το, το εθνικό μας ε, πρόγραμμα δεν είναι ιδιαίτερως ε, φιλικό προς τους νέους, αλλά ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, μια πρωτοβουλία, μια δράση για τους νέους, εξασφαλίζει μια συμμετοχή των νέων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Αλλά όπως σας είπα, δεν υφίσταται τέτοιο πρόγραμμα. Χρειαζόμαστε μηχανισμούς για την ε, ψυχική και σωματική υγεία, για την εξασφάλιση της ψυχικής και σωματικής υγείας και για την δημιουργία καλύτερων επαφών μεταξύ νέων ανθρώπων ως προϋπόθεση για μια βιώσιμη συμμετοχή στην κοινότητα. Και εδώ θα ήθελα να στραφώ προς την προλαλήσα και να πω ότι χρειαζόμαστε ε, νέες προοπτικές ε, διοργανώσεις ή γιορτές ε, σε οποίες θα μπορούν να συμμετάσχουν οι νέοι ε, και να αναπτυχθεί το κοινωνικό κεφάλαιο και ο εθελοντισμός. Και δυνατόν να υπάρξει εναρμόνιση των ε, κρατικών εκπαιδευτικών νόμων αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι συγκεχημένη. Ε, πολλοί ε, έχουν τον τίτλο ε, «Λειτουργεί για τη νεότητα», αλλά αυτό ε, κοινωνική λειτουργία που ασχολούνται με τους νέους, αυτό σημαίνει κάτι άλλο στην κάθε χώρα. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια καλύτερη διαφοροποίηση των διαφόρων εργαλείων όπως Έρικα ε, και Eurodesk εργαλεία τα οποία θέλουμε να διαδώσουμε μεταξύ των νέων ανθρώπων και να τα κάνουμε δημοφιλή. Γιατί τελικά έχει υπάρξει ένα σημείο κορεσμού όπου οι δράσεις μας πάβουν να είναι αποτελεσματικές. Για τα επόμενα δέκα χρόνια λοιπόν χρειαζόμαστε ε, ε, ξεκάθαρα ευρωπαϊκά ήθη, εάν θέλετε, τα οποία θα κινητοποιήσουν ε, τους πολίτες να αισθανθούν ως κομμάτι της μεγάλης ευρωπαϊκής κοινότητας. Για μένα είναι μεγάλη χαρά να ακούω μετά τον εθνικό ύμνο, τον ευρωπαϊκό ύμνο. γιατί έτσι αισθάνεται κανείς ότι συμμετέχει. Είναι μια έκφραση συμμετοχής. Η Βουλγαρία βρίσκεται στα ακραία σύνορα της Ευρώπης, στα εξωτερικά σύνορα μάλλον της Ευρώπης και για μας είναι σημαντική η πρόθεση των σχέσεων μεταξύ γειτονικών χωρών. όσον αφορά τη δημοκρατία και η κοινωνική ένταξη θα πρέπει όλοι να είμαστε από την ίδια πλευρά. Επίσης, σε σχέση γειτονία, ε, γιατί όλα αυτά θα συμβάλλουν στην ειρήνευση. Αυτή τη στιγμή η ειρήνη είναι δεδομένη, αλλά δεν μπορεί να είναι δεδομένη για πάντα. Και τέλος θα ήθελα να απευθυνθώ στους συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ ε, Νεολαίας και το Κίνημα των Προσκόπων, λέγοντας ότι είναι σημαντικό να απευθύνουμε μια έκκληση προς τις χώρες μέλη να χαράξουν, να εκπονήσουν συγκεκριμένα εθνικά προγράμματα δράσης τα οποία θα χτίσουν μια ξεκάθαρη γέφυρα προς την νεολαία της Ευρώπης και έναν ξεκάθαρο μηχανισμό ε, για την υποστήριξη ε, των ε, νέων. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και αναμένω με ανυπομονησία τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ελέγκοβα και θα ξεκινήσουμε και πάλι με την Άλγα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια γρήγορη ερώτηση. Η κυρία Ελέγκοβα αναφέρθηκε ε, επί μακρόν στο θέμα της ένταξης. Μην υπάρχει μια ευρωπαϊκή πολιτική ε, ένταξη, συμπερίληψη, έτσι ώστε αυτέ οι ομάδε νέων που είναι πιο ευάλωτε και που είναι εκτό κοινωνία ε, να μπορέσουν να συμμετάσχουν. Ε, ποια εργαλεία, ποιου μηχανισμού ε, θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε κατά τη γνώμη σα για να προσελκύσουμε ε, ακριβώς τους νέους να συμμετάσχουν στα προγράμματα αυτά. Σε αυτούς που δεν είναι οργανωμένοι ή που αυτή τη στιγμή εν βρίσκονται εκτός. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω το εξής. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή σε εθνικό επίπεδο. Ναι, σε εθνικό επίπεδο μπορούμε να ε, παραδειγματιστούμε από το βουλγαρικό παράδειγμα για να το, μετα... να το μεταφέρουμε ως πλήστη πρακτική σε ευρωπαϊκό. Веднага също ще кажа и това, което се спомена. Не, θα μπορούσα να πω το πώς ε, η οργάνωση των νέων διαμορφώνεται στην ε, Βουλγαρία. Οι περισσότερες οργανώσεις εργάζονται με τον τρόπο αυτό και προσπαθούμε να προχωρήσουμε, αλλά διαπιστώσαμε το εξή. Εάν ε, θέλουμε να εφαρμόσουμε έναν μηχανισμό ελεγγύης στη δική μας εργασία, θα πρέπει να σταθμίσουμε τι δυνατότητες υπάρχουν όσον αφορά την εκπαίδευση και το πώς μπορούμε να συμπεριλάβουμε όλες τις ε, ομάδες ε, νέων δηλαδή να μην υπάρχουν ε, τέλη ή να αποκλείσουμε ή αν το κάνουμε να αποκλείσουμε τις διακρίσεις θα πρέπει να υπάρχει μια καλή προετοιμασία και τις περισσότερες φορές προσπαθούμε να προσελκύσουμε κάποιους εμπειρογνώμονες. Για παράδειγμα, το σύλλογο των κοφών στη Βουλγαρία. Μέσω διερμηνίας στη νοηματική γλώσσα. και έτσι δώσαμε τη δυνατότητα να διαπιστώσουν όλοι ότι υπάρχουν κάποιες αναπηρίες οι οποίες έχουν επιπτώσει στην επικοινωνία. Και αν συνεργαζόμαστε με ανθρώπους που είναι διαφορετικοί, θα έπρεπε αυτό να το λάβουμε υπόψη. Η κυρία Σόντροβα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Ε, δυστυχώς θα πρέπει να πάω στην Επιτροπή Απασχόλησης που έχουμε το θέμα Work-Life Balance. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ελέγκοβα. Είναι το σωστό πρόσωπο, στη θέση. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ε, παρουσιάσετε την εμπειρία σας. Αλλά θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Έτσι όπως βρισκόμαστε όλοι εδώ, όλοι προσπαθούμε οι νέοι άνθρωποι να αποκτήσουν ευκαιρίες για να εκπαιδευτούν, να έχουν ε, πολλές επαφές κλπ. Αυτό είναι το μέλλον Ευρώπη, της Ευρώπης, οι νέοι άνθρωποι. Αλλά θα ήθελα να σας παρακαλέσω και εσείς θα πρέπει να πείτε ότι και εμείς έχουμε κάποιες ε, προσδοκίες από τη δική μας πλευρά. Η Ευρώπη σας χρειάζεται εσάς τους νέους ανθρώπους, και κάνουμε αυτή τη δουλειά ούτως ώστε εσείς οι νέοι άνθρωποι να καταλάβετε την Ευρώπη και να θέλετε μια κοινή ενωμένη Ευρώπη. Ε, αυτό το είπε και ο συνάδελφος, ε, ούτως ώστε να μπορέσετε να επιστρέψετε και πάλι στα, στην πατρίδα σας και να επιστρέψετε αυτό το οποίο σας έχει δωρήσει η Ευρώπη. Αυτή είναι η δική μου εμπειρία και με αυτό θα ήθελα να κλείσω. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν μάλλον ένα statement. Αλλά παρακαλώ κυρία Ελένκεβα. Θα κάνω ένα πολύ σύντομο σχόλιο εδώ. Το πρώτο θέμα του διαφρομένου διαλόγου ήταν το μέλλον της Ευρώπης. Και αυτό ήταν και το βασικό θέμα. Αυτό το οποίο ήρθε από τους νέους ανθρώπους από τη Βουλγαρία, τη Λετωνία και την Αυστρία ήταν το εξής. Ποιος είναι ο ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν στην Ευρώπη. Άρα εστιάζει στην άποψη των νέων ανθρώπων οι οποίοι καλούνται να καθορίσουν το μέλλον τους πράγματι στην Τρόικα αυτή δώσαμε την έμφαση στην επεξεργασία συγκεκριμένων προτάσεων και αυτή θα είναι η επόμενη στόχη των νέων. Το προηγούμενο χρόνο είχαμε τη συζήτηση, είχαμε, ξεκινήσαμε τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, ε, ε, έχουμε πλέον τη Λευκή Βίβλο για το μέλλον της Ευρώπης, αλλά ποιο είναι το καθήκον των νέων της Ευρώπης εδώ. Εγώ είμαι αισιόδοξη γιατί αλλάξαμε το, την αιστεία, την, ε, τον τρόπο που εστιάζουμε τα πράγματα. Ε, κυρία Νέιρα. Θα είμαι σύντομη. Χαίρομαι που επικεντρώνεστε στην κοινωνική ένταξη. Χρησιμοποιείτε όμως τα κοινωνικά μέσα δικτύωση ως πλατφόρμα για να έρθετε σε επαφή με αυτούς τους ε, φοιτητές, τους μαθητές, ε, τους νέους που ζουν σε, στην Ήπεθρο, που είναι ε, αποκλεισμένοι, δεν έχουν εγγυήσει, δεν έχουν πρόσβαση σε δανειοδότηση, δεν θα μπορούσαν άλλωστε να αποπληρώσουν τα δάνεια αυτά. Ε, πώς αντιμετωπίζετε αυτήν την απομόνωση στην Ήπεθρο σε σχέση με αυτούς ε, τους ανθρώπους είναι πολύ στη χώρα μου τουλάχιστον και είναι μια, ένας φαύλος κύκλος. Αν κανείς δεν, δεν ε, ε, πάει προς τους ανθρώπους αυτούς, ε, μένουν οι νέοι άνθρωποι αυτοί εκτός της συζήτησης. Θα πρέπει λοιπόν ε, να υπάρξει χρηματοδότηση έτσι ώστε ε, οι, στις περιοχές αυτές ε, να υπάρξει απαραίτητη στήριξη. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η αποψή σας από αυτού. Η κυρία Λέγκοβα. Η τελευταία συζήτηση κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης στο πλαίσιο του διαδομένου διαλόγου εκεί εκφράσαμε, σε αυτή τη συζήτηση εκφράσαμε τις ανησυχίες μας. Πολλοί άνθρωποι δεν ε, βρίσκονται online και δεν γνωρίζουν τίποτα για τις προσπάθειές μας. Σε εθνικό επίπεδο θα μπορούσα να πω το εξή για τις προσπάθειές μας. Έχουμε εφαρμόσει ένα πολύ πετυχημένο πρόγραμμα με την επωνυμία Ακαδημία γιατί θέλαμε σε κάθε νέο άνθρωπο να δώσουμε την ευκαιρία με την καταβολή κάποιου τέλους για τους συμμετέχοντες και παρέχοντας μια προστασία στους ε, μειονεκτούντες ε, νέους, δημιουργήσαμε ίσες ευκαιρίες. Δηλαδή αποτανθήκαμε στους νέους ανθρώπους και προσπαθήσαμε από κοινού να παρατηρήσουμε το πώς είχαμε μέχρι στιγμής ε, προσλάβει τα πράγματα. Έγιναν κάποιες συνεδριάσεις, προγραμματίσαμε εκδηλώσεις της Ακαδημίας, ήρθαμε σε επαφή με σχολεία και ε, στα μέρη αυτά δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου οργανώσεις νέων. Παρ' όλα αυτά προσπαθήσαμε να απευθυνθούμε σε ακτιβιστές μεταξύ των νέων ώστε να διαδοθούν οι πληροφορίες μας online και offline και προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε τέτοιου είδους ε, κοινότητες ή τόπους όπου ήταν πολύ ισχνές οι, οι δραστηριότητες των νέων. Μετά από αυτή την προσπάθεια στις 13 ε, κοινότητες μπορέσαμε να ε, παρακολουθήσουμε, να διαπιστώσουμε ότι υπήρξε η εξέλιξη κάποιων δραστηριοτήτων και αυτό επιβέωσε την πεποίθησή μας. Δηλαδή μπορούμε να δουλέψουμε στο ψηφιακό επίπεδο, αλλά χρειαζόμαστε και την επιτόπου τη συγκεκριμένη εργασία. Κυρία Ελέγκοβα, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για το πώς θα έχουμε πρόσβαση στους νέους. Πώς όμως θα έρθουμε ε, σε επαφή με εσά, πώς εσείς εργάζεστε ε, σε αυτή την πλατφόρμα, σε αυτό το δομημένο διάλογο, τι μπορούμε να μάθουμε από τη δική σας εμπειρία. Моят, първи младежки обмен беше Η πρώτη μου ανταλλαγή νέων ήταν το 2000-2001. Και θυμάμαι ότι έπρεπε να πάω στη Γαλλία. Είχα το αεροπορικό εισιτήριο, αλλά δεν είχα βίζα και με μεγάλη ανυπομονησία περίμενα τη βίζα μου. Την πήρα πράγμα την τελευταία στιγμή και αυτή ήταν η στιγμή όπου αισθάνθηκα μια τεράστια δυνατότητα ε, να στρατευθώ υπέρ μιας κοινότητας. Τέτοιες δραστηριότητε την εποχή εκείνη δεν ήταν και τόσο δημοφιλείς και ενώ ε, για μένα ε, τέτοιου δουλειά είναι, αποτελεί μεγάλη πηγή έμπνευση και άρχισα να σκέφτομαι, να προβληματίζομαι κατά πόσο υπάρχουν και άλλοι νέοι άνθρωποι σαν και εμένα στη Βουλγαρία και στη συνέχεια ήρθε το πρόγραμμα Νεολαία εν και στο πλαίσιο αυτό διοργανώσαμε μια συνάντηση το 2008 και 2009 με άλλους ε, ε, επικεφαλής τέτοιων ε, κινημάτων και οργανώσεων νέων. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο αύξησε την συνοχή, το βαθμό συνοχής στο εθνικό φόρουμ για την νεολαία. Η επιθυμία μας είναι να δημιουργήσουμε μια καλύτερη Βουλγαρία και μια πιο ελέγγυα Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστούμε. Ο κύριος Μαλίνοφ. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να θέσω την κάπως δυσάρεστη ερώτησή μου στις κύκλους σας γίνονται σκέψεις για το πόσο σημαντικό είναι τουλάχιστον ένα τμήμα των νέων ανθρώπων να μπορεί να παραμείνει στην πατρίδα του και να συμβάλλει στις εκεί εξελίξεις ή δεν υφίσταται για σας αυτό το ερώτημα. Γιατί ε, θα ήθελα να πείτε κάτι για αυτό το θέμα. Όταν εγώ ήμουν ε, νέος, ξεκίνησα τη διατριβή μου με μια υπόθεση. Εσείς ε, καταλήξατε στη δική σας διατριβή σε κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα. Γιατί έχετε εμπειρία σε αυτό το χώρο. Τι θα λέγατε εδώ σχετικά. много е трудно а, да говориш за а, насърчаване или задържане на млади хора όσον αφορά την πρόθεση των νέων ανθρώπων, την, για να μείνουν στην πατρίδα τους, στο χώρο που ξεκίνησαν, αυτή είναι μια πολύ δημοφιλής ρητορία αυτή τη στιγμή στη Βελγαρία γιατί αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο παρατηρώ είναι το εξή. Εάν δούμε τις διαβουλεύσεις για τον ε, διαφορεμένο διάλογο, θα δούμε στο ερωτηματολόγιο συγκεκριμένες ερωτήσεις που αφορούν ε, κάποιες πληροφορίες εν σχέση με το πού ε, χρειάζονται νέοι άνθρωποι. Εάν εξασφαλίσουμε την πρόσβαση στο διαδίκτυο, εάν έχουμε υπηρεσίες που προωθούν τις ε, επαφές μεταξύ νέων ανθρώπων, ε, τα μέρη αυτά, οι ε, τοποθεσίες αυτές θα γινόντουσαν ενδιαφέρουσες για τους νέους ανθρώπους. Εμείς θα παρακολουθήσουμε το πώς διαμορφώνονται αυτά τα αποτελέσματα και στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων θα δούμε πώς ε, νέοι άνθρωποι από όσους συμμετείχαν ε, σε αυτές τις έρευνες ε, πόσοι ανέφεραν ότι δεν θα ήθελαν να πάνε σε μια μεγάλη πόλη λόγω της ρήπανσης και του στρες. Θεωρούν την επιζήμια η διαβίωση στις μεγαλοπόλεις και με τα ψηφιακά εργαλεία θα μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά στο μέρος από το οποίο κατάγονται χωρίς να είναι υποχρεωτικό να πάνε σε μια μεγαλούπολη, ξοδεύοντας εκεί και περισσότερα χρήματα. Τώρα, όσον αφορά την προσωπική διάσταση, θα μπορούσα να απαντήσω προσωπικά στην ερώτησή σας. Ξέρω την θέση της διατριβής μου, η οποία συνδέεται άμεσα με τη σημερινή μου εργασία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι ήταν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανταλλαγή και νομίζω τόσο η Άλγα όσο και οι συντονιστές θα συμπεριλάβουν αυτά τα ερεθίσματα στι εκθέσεις τους. Και θα ήθελα τώρα να ρωτήσω την Επιτροπή κατά πόσο θέλει να πάρει το λόγο. Φαίνεται πως όχι. Άρα θα δώσω στην Άλγα το λόγο για τελικές παρατηρήσεις. Αν έχεις κάποιες τελικές παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Ναι, ήθελα απλά να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές που ήρθαν εδώ να μας εξηγήσουν, να μας παρουσιάσουν συγκεκριμένες ε, καταστάσεις, ε, συγκεκριμένα παραδείγματα. Προετοιμάζουμε εμείς την έκθεση σε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική και έχουμε πολλά να μάθουμε από την μέχρι τώρα πορεία της στρατηγικής και να μπορέσουμε να δώσουμε ένα ε, μήνυμα, να στείλουμε ένα μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ποιο πρέπει να είναι το μέλλον αυτή τη στρατηγική. Σα ευχαριστώ λοιπόν για την ανταλλαγή απόψεων που είχαμε. Ε, χρειάζεται περισσότερη συμμετοχή των νέων στη λήψη αποφάσεων, υποστήριξη στι οργανώσει νεολαία, μια πιο ευρεία ε, πρόσβαση, όχι μόνο οριζόντια, αλλά και σε ό,τι αφορά το, περι, το, περιεχόμενο. Απασχόληση, εκπαίδευση βεβαίω είναι οι κλασικές πολιτικές ε, που αφορούν τους νέους, αλλά ε, και η πολιτιστική ατζέντα, η ψηφιακή ατζέντα, το θέμα της υγείας, ε, είναι πολλά. Δεν θα τα συνοψίσω τώρα. Σας ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ για τις συνεισφορές σας. Σημείωσα όλα αυτά που άκουσα και θα προσπαθήσω να τα συμπεριλάβω σε μια έκθεση πρωτοβουλίας βεβαίως ε, που έχει περιορισμένο εύρος. Δεν μπορούμε δηλαδή να τα συμπεριλάβουμε όλα, θα συμπτύξουμε ό,τι μπορούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Όταν ρώτησα την Επιτροπή, κοίταξα στη λάθος κατεύθυνση και η Επιτροπή βρίσκεται εκεί, κάθεται εκεί και σήκωσε το χέρι. Παρακαλώ, αν επιθυμείτε να πάρετε το λόγο, αλλά όχι περισσότερο από τρία λεπτά. Ναι, είναι όντω σπάνιο ότι να βρεθούμε στο κέντρο εδώ της ομίγυρης είναι και δημιουργεί μια κάποια σύγχυση σε σχέση με τα ε, συνηθισμένα. Ε, σας ευχαριστούμε για την οργάνωση αυτή της ακρόασης. Είναι πραγματικά ενδιαφέρον και για μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εργαζόμαστε σκληρά ε, γύρω την πρότασή μας ε, για να υποβάλουμε μια πρόταση που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες ε, και στις φιλοδοξίες όλων όσων εμπλέκονται στην ατζέντα για τους νέους. Έγινε μια αξιολόγηση της στρατηγικής για τους νέους που επιφέρει κάποια στοιχεία. Είναι σημαντικές πάντως πληροφορίες αυτές. Ε, ε, αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση για την αξιολόγηση, είμαστε έτοιμοι να τη διευκρινίσουμε. Ε, το προηγούμενο έτος είναι ένα έτος ε, όπου αφουγκραστήκαμε τις απόψεις ε, εν ώψη του μέλλοντος της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τους Νέους. Χαιρόμαστε που οι οργανώσεις νέων ε, συνεισέφεραν και αυτές ε, συμμετείχαν ε, μέσω του δομημένου διαλόγου στη συζήτηση αυτή θα παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, τον δομημένο διάλογο και ελπίζουμε να προκύψουν ενδιαφέρουσες ιδέες ο Βίλε αλλά και οι συνάδελφοί του θα μπορέσουν να μοιραστούν περισσότερες πληροφορίες καθώς θα προχωρούμε έχουμε πραγματικά καλές ιδέες και ενδιαφέρουσες που θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε εργαζόμαστε και εμείς σκληρά την πλευρά μας. Ε, αν έχετε να μας ρωτήσετε οτιδήποτε, είμαστε ε, στη διάθεσή σας ε, να μοιραστούμε μαζί σας όλες τις πληροφορίες που έχουμε συλλάξει. Ευχαριστώ πολύ και από τη δική μου πλευρά. Ένα θερμό ευχαριστώ στους ομιλητές μας. Πιστεύω ότι πράγματι ήταν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνεδρίαση. Σε ευχαριστώ πολύ όλους και πιστεύω ότι η διαδικασία που ακολουθήσαμε ήταν κάπως πιο χαλαρή από ό,τι συνήθως. Φαντάζομαι ότι θα μείνουμε σε επαφή, ιδιαίτερα με το Φόρουμ για την Νεολαία, αλλά και με τους άλλους εδώ συμμετέχοντες στο πόντιουμ που έδωσαν σημαντικές επισημάνσεις, αλλά βεβαίως ε, θα ήταν σημαντικό να έχουμε και μια παρακολούθηση της στρατηγικής για την νεολαία. Αλλά βεβαίως, ε, εφόσον πρόκειται για μια στρατηγική είναι σημαντικό να καλέσουμε και εκείνου στους οποίους απευθύνεται η στρατηγική αυτή και νομίζω ότι θα εφαρμόσουμε αυτή την πρακτική στην Επιτροπή μας όπως το κάναμε στο παρελθόν και βεβαίως είμαστε ευγνώμονες για οποιαδήποτε πρόταση, ιδιαίτερα όσον αφορά και την ε, μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση του Εράσμου ΣΥΝ, αλλά και του Σώματος Αλληλεγγύης. Και ελπίζουμε μελλοντικά να λέγεται υπηρεσία αλληλεγγύης. Να παραμείνουμε λοιπόν σε επαφή. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω όλους για το ε, σημαντικό αυτό απόγευμα. Und danke natürlich auch an unsere Dolmetscherin dafür, dass sie uns wie immer hilfreich zur Seite gestanden haben. Die nächste Sitzung findet statt am 21. Η επόμενη συνεδρίαση θα είναι στις 21 Φεβρουαρίου από 9 ως 12.30 και από 2.30 ως 6 και την 5η στις 22 Φεβρουαρίου από τις 9 ως τις 12.30. Έως τότε, καλό βράδυ.